Παπα-Νικολάου, <laughs> δεν είσαι σοσιαλιστής, γιατί κάθεσαι με τους σοσιαλιστάς. Έλα από εδώ παρακαλώ. Όχι και τέτοια ευελιξία, βρε παιδιά. Λοιπόν, σας καλωσορίζω όλους. Ευχαριστώ πολύ που προσήλθατε σήμερα. Δυστυχώς είχαμε πολύ μεγάλο διάλειμμα από τις 11 μέχρι τώρα και μερικοί φαίνεται εντωμεταξύ εξαφανίστηκαν. Αλλά χαίρομαι που μπορούμε να συναντήσουμε τον Υπουργό Παιδείας της Ελληνικής Προεδρίας. Παιδείας και θρησκευμάτων βλέπω εδώ, τον κύριο Αρβανιτόπουλο. Σας καλωσορίζω λοιπόν και σας και το προσωπικό σας και θα σας δώσουμε αμέσως το λόγο για να μας πείτε τι φρονείτε για τους επόμενους μήνες. Δεν είναι πάρα πολύ καιρό, δεν θα αλλάξετε τον κόσμο ούτε εσείς ούτε εγώ σε έξι μήνες, αλλά αφού μιλήσατε, συνεννοηθήκατε με τη Λιθουανική Προεδρία και με την επόμενη, νομίζω ότι θα μπορέσετε να μας πείτε ποιες είναι οι προτεραιότητες σας. Ορίστε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, είναι μεγάλη τιμή για μένα η παρουσία μου και ελπίζω να μην είναι αλήθεια το νέο που άκουσα ότι θα φύγετε, δεν θα είστε υποψήφια στην επόμενη θητεία. Σε αυτή την περίπτωση θέλω να σας συγχαρώ για την καριέρα σας και για όλες σας τις επιτυχίες όπως το Erasmus Συν που είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της και σας ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι Ευρωβουλευτές, έχω την ιδιαίτερη τιμή και χαρά να βρίσκομαι σήμερα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να σας παρουσιάσω τις προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας και θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω επισημένοντας ότι η παιδεία αποτελεί το θεμέλιο των προσδοκιών μας για ένα συλλογικό μέλλον με γνώμονα την αρμονική συμβίωση αλλά και την προαγωγή των ευρωπαϊκών αξιών. Παράλληλα όμως, η παιδεία οφείλει να δίνει στους νέους μας τις δεξιότητες αλλά και τις ικανότητες για τη βελτίωση της προβασιμότητάς τους στην αγορά εργασίας. Γι' αυτό σε αυτή τη βάση η ελληνική προεδρία καλείται σε συνεργασία με όλα τα κράτη μέλη με το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο με την ευρωπαϊκή επιτροπή να προωθήσει την υλοποίηση των στόχων της ευρωπαϊκής ένωσης. Κυρίες και κύριοι, το σύγχρονο σχολείο αντιμετωπίζει σήμερα θεμελιώδη διλήμματα που αφορούν τόσο το επίπεδο του περιεχομένου και της ποιότητας της παρεχόμενης γνώσης, όσο και το επίπεδο της οργανωτικής δομής της λειτουργίας του, και ειδικότερα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο παγκόσμιας κοινωνικής και οικονομικής κρίσης. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η σημερινή ανάγκη προσδιορίζεται στη δημιουργία μιας κουλτούρας μάθησης η οποία θα δίνει έμφαση σε μια μακρόπνοη και συνεχή μαθησιακή διαδικασία που θα ξεκινάει από την προσχολική ηλικία έως και την τρίτη ηλικία και θα καλύπτει κάθε μορφής εκπαίδευση και κατάρτιση που θα διέπεται βέβαια από τις ουμανιστικές αρχές της κοινωνικής ισοτιμίας, της κοινωνικής συνοχής. Παρά τα ενθαρρυντικά σημάδια της σταδιακής ανάκαμψης στην Ευρώπη, όλοι γνωρίζουμε ότι πολλά απομένουν να γίνουν, προκειμένου να αντιστραφούν πλήρως οι επιπτώσεις της κρίσης, η οποία έχει πλήξει κέρια ιδιαίτερα τους νέους ανθρώπους, μια ιδιαίτερα ευάλωτη κατηγορία του ενεργού πληθυσμού, με μέσο ποσοστό της ανεργίας στους νέους να φτάνει στο 23%, 23,5% αλλά και με χώρες να παρουσιάζουν ποσοστά ανεργίας στους νέους πάνω από το 50%. Όπως για παράδειγμα η χώρα μου. Παράλληλα το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας εμφανίζεται σε άτομα με λυπείς δεξιότητες. Και εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ένα 20% του ενεργού πληθυσμού παρουσιάζει χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων και κατανόησης μαθηματικών υπολογισμών, ενώ ένα 25% δεν διαθέτει τις απαραίτητες δεξιότητες για να κάνει αποτελεσματική χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας. Καλούμεθα λοιπόν τα κράτη-μέλη να αντιμετωπίσουμε μια κρίσιμη δέσμη ζητημάτων για το μέλλον της ευρωπαϊκής εκπαίδευσης με στόχο την αντιμετώπιση της διπλής πρόκλησης της νεανικής ανεργίας αλλά και του ελλείμματος δεξιοτήτων διατηρώντα βέβαια πάντοτε στην εκπαιδευτική μας διαδικασία τον ουμανιστικό της χαρακτήρα. Σε αυτό το πλαίσιο, οι προτεραιότητες της ελληνικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την νεολαία διαρθρώνονται στους εξή θεματικούς πυλώνες. Πρώτον, η διασφάλιση της ποιότητας σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Δεύτερον, αποτελεσματική και καινοτόμος εκπαίδευση και κατάρτιση τρίτον κοινωνική συνοχή και τέταρτον η επιχειρηματικότητα των νέων. Όσον αφορά τη διασφάλιση της ποιότητας σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης, γνωρίζουμε ότι η εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα εξαρτάται πρωτίστως από τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας παρεχομένων γνώσεων και δεξιοτήτων. Και αυτό και η πρώτη μας προτεραιότητα εστιάζεται ακριβώς αυτό, στη διασφάλιση της ποιότητας σε όλα τα επίπεδα κάτι που θα μας επιτρέψει σε όλα τα κράτη-μέλη και στην Ευρώπη συνολικά να υπερβούμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, να διατηρήσουμε την, ανταγωνιστικότητά μας και η Ευρώπη βέβαια να διατηρήσει τη θέση της σε έναν πρωταρχικό, σημαντικό πρωταγωνιστή στο διεθνές στερέο. Η διασφάλιση της ποιότητας στην εκπαίδευση απαιτεί την ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων, καινοτόμων εργαλείων και μέσων. Και στο πλαίσιο αυτή της προσπάθειας είναι ιδιαίτερα σημαντική η κατάλληλη εκπαίδευση των εκπαιδευτικών μας για την προώθηση νέων δεξιοτήτων, για την εφαρμογή νέων καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας. Γιατί χωρίς αμφιβολία ο ρόλος τους είναι κρίσιμος. Με το θέμα αυτό έχει ήδη ασχοληθεί το Συμβούλιο 2009 με συμπεράσματα για την επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας υπήρξε συζήτηση για το ρόλο του εκπαιδευτικού, ενώ πρόσφατα η Λιθουανική Προεδρία υιοθέτησε συμπεράσματα για την ηγεσία της εκπαίδευσης, για τα ηγετικά στελέχη της εκπαίδευσης. Εμείς θα κλείσουμε τον κύκλο αυτών των συζητήσεων, του σημαντικού αυτού θέματος, της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, λαμβάνοντας βέβαια πάντοτε υπόψη τις σύνθετες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν κατά την άσκηση του λειτουργήματός τους. Παρότι όμω υπάρχουν πολιτικέ υποστήριξη των εκπαιδευτικών αλλά και των σχολικών διευθυντών σε ορισμένα κράτη-μέλη, πολύ συχνά βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν συγκροτημένε πολιτικέ ή ρυθμίσει για του τρόπου επιλογή των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών του, δεν υπάρχουν συγκροτημένε πολιτικέ για τα απαιτούμενα προσόντα ή για την οργάνωση τη διαρκού επαγγελματική του εξέλιξη. Η προσέγγιση μας θα υιοθετήσει τους στόχους που αναδείχθηκαν στο συνέδριο Ένταξη, Καινοτομία και Βελτίωση, η επαγγελματική ταυτότητα των εκπαιδευτών, που διοργανώθηκε από την Ιρλανδική Προεδρία στις 18 και 19 Φεβρουαρίου. Στόχοι όπως ο επανασχεδιασμός της διαδικασίας πρόσληψης και επιλογής των καλύτερων εκπαιδευτικών, η αποτελεσματικότερη εισαγωγική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, η συστηματική υποστήριξη στα πρώτα βήματα της επαγγελματικής τους πορείας, η συνεργατική επαγγελματική μάθηση, η ανατροφοδότηση των εκπαιδευτικών, ο προσδιορισμός των ικανοτήτων που απαιτούν οι εκπαιδευτές των εκπαιδευτικών και ούτω καθεξής. Η εκπαίδευση των εκπαιδευτών μας, των εκπαιδευτικών μας, είναι ένα μείζον ζήτημα εκπαιδευτικής πολιτικής και επενδύει στο μέλλον της παιδείας και στη νέα γνώση. Γι' αυτό θα εργαστούμε από κοινού με τους εταίρους μας για την προώθηση συμπερασμάτων, για τη διασφάλιση της ποιότητας σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευση και κατάρτισης, καθώς και τα δύο αυτά θέματα είναι αλληλοσυνδεόμενα και αλληλοσυμπληρούμενα. Η δεύτερη προτεραιότητα είναι η εγγύηση συνθηκών αποτελεσματικότητας, εξωστρέφειας, κινητικότητας και απασχολησιμότητας. Με κύριους πυλώνες την διαρκή και καινοτόμο επένδυση στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση. Όλοι γνωρίζουμε ότι σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία της γνώσης που συναρτάται ολοένα και περισσότερο με την ανάπτυξη πολλαπλών δεξιοτήτων, πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να προσφέρουμε αποτελεσματική εκπαίδευση η οποία θα συνάδει με την ανάπτυξη, με τα ζητούμενα από την αγορά, με θέματα ανταγωνιστικότητας. Και βλέπουμε ότι η Ελληνική Προεδρία συμπίπτει με την έναρξη ενό πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου, στο οποίο περιλαμβάνεται το νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+, και η νέα γενιά διαρθωτικών και επενδυτικών ταμείων, τα οποία βέβαια είναι επιτακτικό να επενδύσουν στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Υπάρχει μια μεγάλη ανάγκη για υποστήριξη μακροχρόνιας επένδυσης, για επικέντρωση στις ανισότητες, για προσέλκυση, εκπαίδευση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών, των διευθυντών σχολείων, των εκπαιδευτών των εκπαιδευτικών, καθώς βέβαια και υποστήριξη της ανάπτυξης των ανοιχτών εκπαιδευτικών μέσων και των ανοιχτών μαζικών διαδικτυακών μαθημάτων. Βλέπουμε όλοι ότι οι νέες εξελίξεις έχουν αυξήσει δραματικά τις ευκαιρίες μάθησης. Οι ανοιχτές τεχνολογίες έχουν τη δυνατότητα να επιτρέπουν στα άτομα να μαθαίνουν οπουδήποτε, οποτεδήποτε, μέσω οποιασδήποτε συσκευής, με την υποστήριξη οποιοδήποτε. Η ανάδυση αυτών των καινοτόμων μοντέλων για τη διδασκαλία και τη μάθηση όπως τα ανοιχτά μαζικά διαδικτυακά μαθήματα, τα περίφημα MOOCs, θα μεταμορφώσουν την εκπαίδευση, είναι σίγουρο. Και θα δημιουργήσουν ένα νέο ανταγωνισμό και κέντρα αριστείας σε όλο τον κόσμο. Αυτή η διεθνοποίηση της εκπαίδευσης, είτε επειδή οι σπουδαστές αναπτύσσουν μεγαλύτερη κινητικότητα, είτε επειδή οι πάροχοι της εκπαίδευσης και κατάρτισης προσφέρουν υπηρεσίες σε περισσότερες της μίας χώρας, συμβάλλουν ακόμα περισσότερο στη διεύρυνση της εκπαιδευτικής προσφοράς. Γι' αυτό υποστηρίζουμε την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το άνοιγμα της εκπαίδευσης, Opening Up Education, με έμφαση στην ενίσχυση του διαλόγου γύρω από τις ψηφιακές δεξιότητες. Πρόκειται για μια αναγκαία, κατά την άποψή μας, πρωτοβουλία, αφού οι προβλέψεις κάνουν λόγο ότι το 90% των θέσεων εργασίας στο μέλλον θα απαιτούν κατελάχιστο κάποιες βασικές ψηφιακές δυνατότητες και δεξιότητες. Και στις μέρες μας γνωρίζουμε ότι μόνο το 25% των μαθητών ηλικίας 9 ετών φοιτούν σε σχολεία, μαθητεύουν σε σχολεία με υψηλές ψηφιακές υποδομές και προδιαγραφές, ενώ παραπάνω από το 50% των μαθητών στα κράτη-μέλη ακόμα και σήμερα μπορεί να μην κάνουν χρήση καθόλου ψηφιακών εγχειριδίων ή άλλων ψηφιακών εκπαιδευτικών μέσων. Αυτό πρέπει να το αλλάξουμε. Και παράλληλα βέβαια θα πρέπει να επιλύσουμε άμεσα τα νέα ζητήματα που αναφύονται, ζητήματα δηλαδή διασφάλισης της ποιότητας, των πνευματικών δικαιωμάτων και το θέμα της προσβασιμότητας σε αυτά τα μέσα από όλους. Παράλληλα θα μας απασχολήσει το ζήτημα του δίκτυα αναφοράς για τη γλωσσομάθεια, το Language Benchmark. Μια δράση η οποία συνεπικουρεί το στόχο της αποτελεσματικότητας αλλά και της διασφάλισης ποιότητας. Γιατί οι γλωσσικές ικανότητες θεωρούνται και είναι δεξιότητες κλειδιά οι οποίες διευκολύνουν την κινητικότητα, βελτιώνουν την προσβασιμότητα των Ευρωπαίων πολιτών στην αγορά εργασίας και διευκολύνουν τον πολυπολιτισμικό διάλογο. Και ιδιαίτερα στο τρέχον αυτό περιβάλλον, η βελτιωμένη, το οικονομικό αυτό περιβάλλον που ζούμε, η βελτιωμένη διδασκαλία αλλά και η εκμάθηση αρκετών γλωσσών είναι πολύ σημαντική. Γνωρίζουμε ότι σε συνέχεια του αιτήματο του Συμβουλίου και των αποτελεσμάτων τη Ευρωπαϊκή Έρευνα για τι Γλωσσικέ Δεξιότητε, η Επιτροπή διατύπωσε μια πρόταση για έναν ευρωπαϊκό δίκτυο αναφορά γλωσσών στην επικοινωνία του 2012, αναθεωρώντας την εκπαίδευση, σύμφωνα με τον οποίο μέχρι το 2020 το 50% των 15χρονων μαθητών θα πρέπει να κατέχουν το επίπεδο του ανεξάρτητου χρήστη της πρώτης ξένης γλώσσας και τουλάχιστον το 75% των μαθητών του γυμνασίου να διδάσκονται μια δεύτερη ξένη γλώσσα. Νομίζω ότι ένας ευρωπαϊκός δείκτης αναφοράς μπορεί να επιτρέψει την ανάπτυξη ευρωπαϊκών υποστηρικτικών μέτρων και εθνικών πολιτικών στη βάση αποτελεσμάτων παρακολούθησης και κατά συνέπεια να βοηθήσει τις εθνικές πολιτικές να αξιοποιήσουν και να αξιολογήσουν τις επενδύσεις του σχολικού συστήματος στην διδασκαλία ξένων γλωσσών. Στον τομέα της νεολαίας, η ελληνική προεδρία στο πλαίσιο της κοινωνικής ένταξης των νέων, η οποία αποτελεί μια θεματική προτεραιότητα του τρίου, στοχεύει στην αντιμετώπιση του φαινομένου του κοινωνικού αποκλεισμού των νέων. Σύμφωνα με την στρατηγική Ευρώπη 2020 θα ασχοληθούμε και θα προσπαθήσουμε να προωθήσουμε στο Συμβούλιο συμπεράσματα για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των νέων, δίνοντας έμφαση στην κοινωνική επιχειρηματικότητα και την επιχειρηματικότητα στον τομέα του πολιτισμού. Και επίσης θα προσπαθήσουμε να προωθήσουμε ψήφισμα στο Συμβούλιο για τον διαρθρωμένο διάλογο με τους νέους, για την ενίσχυση της κοινωνικής ενσωμάτωσης. Στόχος είναι να διευρύνουμε και να εμβαθύνουμε τη διαδικασία του διαρθρωμένου διαλόγου, έτσι ώστε όλοι οι νέοι ανεξαιρέτως να εμπλακούν σε αυτή τη διαδικασία. Και βεβαίως να ενθαρρύνουμε τον διάλογο μεταξύ των κρατών μελών για τις θεματικές προτεραιότητες του προγράμματος εργασιών στον τομέα της νεολαίας. Τέλος, στο πλαίσιο της Προεδρίας θα γίνουν αρκετά συνέδρια συνέδρια που θα αφορούν την προσχολική αγωγή, συνέδρια που θα αφορούν την αναντιστοιχία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης δεξιοτήτων των συστημάτων εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας, συνέδριο που θα αφορά το νέο σύστημα κατάταξης των πανεπιστημίων, το U Multirank, καθώς και την Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νεολαίας. Και θα είναι μεγάλη μας τιμή να παρευρεθείτε σε αυτά τα συνέδρια και φυσικά είστε ευπρόσδεκτοι της Προεδρίας σε αυτά τα συνέδρια. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, ευρωβουλευτές, η παιδεία συνιστά τον διάβλο για την αναζήτηση, την θεμελίωση και την μετάδοση της γνώσης. Την πιο ουσιώδη και ανταποδοτική επένδυση στους νέους με όρους κοινωνικής συνοχής, αλλά και επιστημονικής και επαγγελματική εξέλιξης. Είναι, θα λέγαμε, και το οξυγόνο της Ευρώπης ως κοινότητα σκεπτομένων και υπεύθυνων πολιτών ικανών να αναμετρηθούν με τις νέες προκλήσεις σε ένα ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον. Η παιδεία θα έλεγα ότι αναζωογονεί και, την, το ίδιο το ευρωπαϊκό ιδεώδες για τη διάπλαση μιας Ευρώπης ικανής να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις με όραμα, με σχέδιο, με αλληλεγγύη, ιδιαίτερα σε αυτές τις περιόδους της δύσκολης κρίσης που διερχόμεθα. Θα ήθελα λοιπόν να εκφράσω εκ μέρους της Ελληνικής Προεδρίας τις θερμές ευχαριστίες μας στην Ιρλανδική και την Λιθουανική Προεδρία, σε όλους τους εταίρους, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συνεργασία κατά την περίοδο της προετοιμασίας που προηγήθηκε και που είμαι σίγουρος ότι θα συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της Προεδρίας και να διαβεβαιώσω ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε από την ε, πλευρά μας σε αυτόν τον περιορισμένο χρόνο της Προεδρίας για να συμβάλλουμε στους κοινού στόχους, τους ευρωπαϊκούς στόχους, στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας. Για μια Ευρώπη της μάθησης, των, της γνώσης και των αξιών. Σας ευχαριστώ. Vielen Dank, Herr Minister. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Στο Συμβούλιο Υπουργών έχω την εντύπωση ότι σωστά σκέπτονται για την εκπαίδευση και την κατάρτιση και αν η σκέψη ακολουθηθεί και από πράξεις τότε όλοι θα χαρούμε ιδιαίτερα. Χτες και σήμερα μιλάγαμε για τις νέες τεχνολογίες και τους ανοιχτούς εκπαιδευτικούς πόρους. Ο συνάδελφος Ιβάν ήταν ο, είναι ο εισηγητής, είχαμε και εμπειρογνώμονες καλεσμένους χτες που έκαναν τις προτάσεις τους και αν έχουμε και εσάς στο πλευρό μας τότε θα έχουμε κάποιον στο Συμβούλιο που φροντίζει οι προτάσεις να συζητούνται και οι συνάδελφοί σας από τις διάφορες χώρες θα προσπαθήσουν και εκείνοι να ακολουθήσουν τις συστάσεις Μόνο αν πάρουμε στα σοβαρά όλα αυτά που είπαμε σήμερα θα πετύχουμε τους στόχους που αναφέρατε κι εσείς και που τους συζητούσαμε και εμείς χθες και σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη συνεργασία σας με τη Λιθουανική Προεδρία και την Ιρλανδική για το, στα πλαίσια του έρασμου ΣΥΝ. Νομίζω ότι χρειάστηκαν πολλές προσπάθειες και από την πλευρά του Συμβουλίου ώστε να δοθούν οι διαβεβαιώσεις που χρειάζεται το Κοινοβούλιο για να τα αποδεχτεί όλα αυτά. Και νομίζω ότι καταρτήσαμε από κοινού ένα εξαιρετικό κείμενο. Ελπίζομαι ότι θα το εφαρμόσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως πρέπει. Η Μαρή Τερές Σάντζε Σμίθ ζήτησε πρώτη το λόγο. Αρχίζει η συζήτηση. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε ιδιαίτερα. Συμφωνώ απόλυτα με όσα υπόθηκαν ε, Δίκιο έχετε η προτεραιότητα της ελληνικής προεδρίας για την παιδεία, την κατάρτιση, την εκπαίδευση. Αν αποδώσει καρπούς, τότε θα συμφωνούσαμε σίγουρα για δύο λόγους. Η ανεργία είναι ιδιαίτερα υψηλή, αφορά κυρίως τους νέους και διαπιστώνουμε καθημερινά ένα ευροσκεπτικισμό από τα περισσότερα κράτη της Ευρώπης. Άρα λοιπόν ο ρόλος της παιδείας είναι σημαντικότατος για να δώσουμε τη μάχη μας κατά των δύο αυτών δεινών που πλήττουν σήμερα την Ευρώπη. Κατανοούμε τις οικονομικές δυσκολίες της Ελλάδος και άλλων χωρών του Νότου αλλά και της Γαλλίας Έχουμε δύσκολες καταστάσεις, έχουμε τουλάχιστον 25% ανεργία στους νέους, χρειάζεται λοιπόν να δώσουμε τη μάχη μας, ένα αγώνα κατά της δυσκολίας αυτής. Η παιδεία και εγώ είμαι εκπαιδευτικός όπως και ο πρόεδρος, όπως και ορισμένοι άλλοι από μας. Και το κλειδί εκεί είναι στην εκπαίδευση, στην κατάρτιση που πρέπει να ξεκινάει από πολύ νεαρή, τρυφερή ηλικία και πολλοί κόσμος που είναι απελπισμένος είναι εύκολη λία για τα άκρατα πολιτικά. Και τώρα αναλαμβάνει την Προεδρία τη στιγμή αυτή που ε, ξεκινάμε και με τον προϋπολογισμό μας και με ορισμένα προγράμματα πολύ σημαντικά για την νεολαία στην Επιτροπή μας. Ο έρασμος, το έρασμο ας πούμε και άκουσα την κινητικότητα και διάφορες άλλες λέξεις που ακριβώς έχουν να κάνουν με τα προγράμματα αυτά. Και περιμένουμε όλοι μας να δούμε τι θα κάνουν τα κράτη, πώς θα τα προωθήσουν αυτά τα προγράμματα και πόσο γρήγορα θα ασχοληθούν με τους νέους. Γιατί πολλές φορές στην Ευρώπη μας κατηγορούν για καθυστέρηση, για αργοπορία. Θα πρέπει να δείξουμε ε, ότι αυτά που είπαμε στην σύνταξη αυτών των προγραμμάτων τα εφαρμόζουμε για την απλοποίηση, για την αποτελεσματικότητα που επιθυμούμε και όλα αυτά θα πρέπει σήμερα να είναι ορατά. Και από την Προεδρία σας βέβαια, γιατί είναι μια Προεδρία που τώρα ξεκινάει με προγράμματα, αλλά και η Προεδρία λίγο πριν ε, την, ε, τις ευρωεκλογές, την ανέωση της θητείας των διαφόρων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και υπενθυμίζω ότι το είπατε ότι τα διαρχωτικά ταμεία θα πρέπει να βοηθήσουν την εκπαίδευση γιατί έχουν καινούρια μέσα, διαθέτουν καινούρια μέσα και εγώ από την ομάδα μου, το πολιτικό μου κόμμα για τον κανονισμό κλπ. Ε, ήμουν η αρμόδια και θα πρέπει όλα αυτά να είναι στην εκπαίδευση, στην κατάρτιση και το, κυρίως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με σημαντικές πιστώσεις ε, και μέσα παραπάνω από ό,τι μπορούμε να υπολογίζουμε πάρα πολλά χρήματα και να βοηθηθεί έτσι και η παλαιματική κατάρτιση που αποδίδεται σημασία σήμερα περισσότερο καμιά φορά και από την πανεπιστημιακή και να πρέπει να βρούμε και μια συνεργασία ανάμεσα στον επιχειρηματικό κόσμο, μια συμμαχία και στην εκπαίδευση και έτσι η εκπαίδευση που θα παροτρύνουμε να δημιουργήσει θέσεις εργασίας και περιμένουμε ε, και νέους αριθμούς και θα πρέπει να κερδίσουμε τη μάχη μας κατά της ανεργίας η Ντόρις μίλησε για όσα είπαμε χθε εδώ, το e-learning ας πούμε και τα MOOC και εκεί είναι το μέλλον. Μέσα σε αυτά τα μέσα εκμάθησης θα πρέπει να διαθέτουμε κάθε μέσο για μια πρόσβαση και στη νέα τεχνολογία ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την κατάρτιση. Σίγουρα υπάρχει μια κάποια καθυστέρηση εργοπορία γιατί δεν είναι ακόμα έτοιμοι να χρησιμοποιήσουν αυτές τις τεχνολογίες. Άρα λοιπόν σίγουρα θα αποτελέσουν μέσα εργαλεία για τις νέες μεθόδους εκμάθησης αλλά ταυτόχρονα θα έχουν πρόσβαση όλοι ανεξαρτήτου ηλικίας σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους για την κατάρτισή τους. Δυστυχώς διακόπτεται το μικρόφωνο της ομιλήτριας, δεν την ακούμε. Διακόπτεται και πάλι. Κλείνει το μικρόφωνο της ομιλήτριας. Εντάξει, ναι, ναι. Λειτουργεί τώρα. Λοιπόν, Άλλο ένα στοιχείο αναφέρεται σημαντικό για την κινητικότητα, την αναγνώριση των προσόντων, των δεξιοτήτων, των επαγγελματικών και κυρίως αυτές που έχουν, αυτά που θα έχουν σχέση με τις νέες τεχνολογίες και επειδή είμαι εκπαιδευτικό ήδη και διαπιστώνω ότι η κατάρτιση των εκπαιδευτικών ε, και από τις κυβερνήσεις ε, τους ενδιαφέρει αλλά ακόμα δεν βρήκαμε το μαγικό ραβδάκι, τη μαγική μέθοδο θα πρέπει να παροτρύνουμε τα κράτη-μέλη να αφιερώσουν και χρόνο και μέσα αλλά ταυτόχρονα μια κάποια εναρμόνιση να σημειωθεί ανάμεσα στα διάφορα συστήματα στην Ευρώπη, γιατί έτσι θα ξαναβρούμε την υγεία μας μέσω αυτών των προτεραιοτήτων. Ευχαριστούμε Μαρή Η κυρία Παλιαδέλη. Σωρίσω στα ελληνικά κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ που είστε εδώ. Καλή επιτυχία στο εξάμεινο, που δεν είναι εξάμεινο, είναι ε, ομολογώ ότι διάβασα τις ε, προτάσεις σας και μας βρίσκεται από ό,τι ξέρω τους περισσότερους σύμφωνους. Καταλαβαίνω βέβαια τις δυσκολίες στην εφαρμογή τους. Θα είμαι πολύ σύντομη, ξεκινώντας με μια παρατήρηση που ενδεχομένως αφορά την Κομισιόν και όχι εσάς, αλλά ίσως μπορείτε να κάνετε κάτι. Ε, το Erasmus Plus, για το οποίο ε, δουλέψαμε πάρα πολύ και σε αυτή την Επιτροπή και στο Κοινοβούλιο, δυστυχώς δεν έχει μεταφραστεί ακόμη σε άλλες γλώσσες εκτός από, το, αγγλικό κείμενο. Επομένως, ε, ξέρω καλά ότι το ελληνικό Ίδρυμα ε, Κρατικών Υποτροφιών το μεταφράζει μόνο του. Θα φροντίσετε να πιέσετε την Κομισιόν να ε, προχωρήσει τη μετάφραση όλων των επίσημων γλωσσών της Ένωσης. συμφωνώ απόλυτα με την ανάγκη για την, ανάγκη της διεθνοποίησης των πανεπιστημίων. Θα ήθελα εδώ να επισημάνω ε, μια, έναν κίνδυνο που προκύπτει από την κρίση και ενδεχομένως και από την άποψη ότι θα βγούμε από αυτήν μόνο αν είμαστε έτοιμοι και, ε, να, να ανταποκριθούμε σε κριτήρια όμως τα οποία ξεχνούν το παρελθόν μας. Η Ευρώπη είναι η μητέρα των επιστημών ε, και οι ανθρωπιστικές επιστήμες δυστυχώς μαράζουν συνεχώς. Θα πρότεινα λοιπόν ότι μία προσπάθεια για την διατήρησή τους και στο επίπεδο της θεωρίας και στο επίπεδο της έρευνας για το οποίο κάναμε προσπάθειες εδώ στο Κοινοβούλιο που δυστυχώς όμως δεν κατέληξαν εκεί που θα θέλαμε αν δηλαδή μια πρόταση δική σας ε, στο Συμβούλιο ε, προκειμένου να δώσει την εντολή στην Κομισιόν να συντάξει ένα κείμενο που να αφορά στους τρόπους με τους οποίους θα διατηρηθούν οι ανθρωπιστικές επιστήμες και θα υποστηριχτεί η έρευνά τους θα ήταν πραγματικά πολύτιμη συμβολή για μια Ευρώπη που θέλουμε να κρατήσουμε ε, και τις, τις οποίες τις αρχές θέλουμε να κρατήσουμε. Και μια τρίτη ερώτηση. Πώς, ε, ελπίζετε ότι με τις, με περικοπές ε, στα κονδύλια για την εκπαίδευση κάτι που προκύπτει από την τεράστια οικονομική κρίση που βιώνουν κυρίως οι χώρες της, του Νότου μπορούμε να εφαρμόσουμε τέτοια φιλόδοξα προγράμματα σαν αυτά που ε, προτείνονται μέσα από το Erasmus 3 και τα οποία αισιοδοξείτε να υποστηρίξετε. Ευχαριστώ πολύ. Äh, Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπόρις. Ε, Καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσίασή σας, αλλά πρέπει να σας πω ότι και πρέπει να σας πω ότι όλα όσα μας είπατε μας καθησυχάζουν ως προς τους στόχους σας για την παιδεία και τη χρησιμοποίηση, όπως είπατε, όλων των δυνατοτήτων που υπάρχουν μεταξύ των οποίων και τις νέες τεχνολογίες. Πολύ σημαντικό και για την παιδεία. Οι άξονες που αναφέρατε, οι προτεραιότητες, με στόχο την καλύτερη, τη μεγαλύτερη καταπολέμηση της ανεργίας των νέων είναι πολύ σημαντική και εμείς έχουμε μιλήσει για αυτά τα θέματα συχνά, για τον προϋπολογισμό, αλλά ο βαθμός μεταφοράς της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας στα κράτη-μέλη διαφέρει από το ένα στο άλλο. Και βέβαια η ανάλυση πρέπει να γίνει ένα-ένα ε, κράτος. Θα θέλαμε όμως να είστε ο συνομιλητής μας εδώ στο Κοινοβούλιο ως εκπρόσωπος της Προεδρίας. Έχουμε πολλούς πόρους που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να επιταχυνθεί η διαδικασία της ηλεκτρονικής μάθησης. Ο έρασμος ήταν μεγάλη επιτυχία και οι αρμόδιοι εισηγητές μας εδώ γνωρίζουν τι αγώνα κάναμε γι' αυτό. Και πετύχαμε 50% αύξηση των κοντιλίων για τα επόμενα χρόνια, αν και συνολικά περικόπηκε ο προπολογισμό. Το θέμα λοιπόν τώρα είναι πώς θα χρησιμοποιηθούν τα διαθέσιμα χρήματα και ποια θέματα θα προωθηθούν. Έχουμε πάνω από 15 δισεκατομμύρια αυτή τη φορά στον έρασμο. Πρέπει να δούμε πώς θα γίνει καλύτερη δυνατή χρησιμοποίηση και να μάθουν περί εράσμου όλοι οι φοιτητέ. Υπάρχουν δυνατότητες αλλά πρέπει και να μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε και να τις εκμεταλλευτούμε. Όσο για την επαγγελματική εκπαίδευση υπάρχει το γερμανικό παράδειγμα που είναι πολύ θετικό. Η ανεργία των νέων με αυτό θα καταπολεμηθεί. Το θέμα δεν είναι μόνο να διορθωθεί η οικονομία αλλά να είναι ισχυρό και το σύστημα, το εκπαιδευτικό σύστημα που θα επιτρέψει στους νέους να μπουν στην αγορά εργασίας. Είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε ότι η φωνή σας και η φωνή των άλλων υπουργών πρέπει να ακουστεί. Πρέπει να τονίσουμε ότι αξίζει τον κόπο να επενδύουμε και στις δεξιότητες των καθηγητών των εκπαιδευτικών, ιδιαίτερα ως προς τις νέες τεχνολογίες. Πρέπει να προετοιμαστούν και οι εκπαιδευτικοί για αυτό το θέμα για να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν τις νέες ευκαιρίες και επομένως να αυξήσουν και αυτοί τις δεξιότητες τους. Ξέρουμε ότι οι Υπουργοί Παιδείας δεν χρησιμοποιούν πάντοτε, δεν γνωρίζουν πάντοτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο πώς θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν τα ευρωπαϊκά χρήματα καλύτερα και εσείς θα ήσασταν ο καταλληλότερος για να το διαδώσετε αυτό θα γίνει μια νέα καμπάνια πληροφόρησης, πρέπει να γίνει, για την καλύτερη επαναλαμβάνω δυνατή χρηματοδότηση των υπαρχών κονδυλίων. Ευχαριστούμε. Ο η, κυρία Παλια... η κυρία Κοπά είναι η τελευταία που θα λάβει το λόγο σε αυτό το γύρο. Όχι κυρία Παλιαδέλη, κυρία Κοπά. Τορίσουμε με τη σειρά μου τον Υπουργό. Είναι μεγάλη χαρά που τον έχουμε εδώ και να ευχηθώ από την καρδιά μου τα καλύτερα για την ελληνική προεδρία ειδικά σε αυτό τον πολύ κρίσιμο τομέα. Κύριε Υπουργέ, το μεγάλο πρόβλημα των νέων στην Ευρώπη, όπως πολύ σωστά επισημάνατε, είναι η νεανική ανεργία. Στη χώρα μας ξεπερνάει το 62% παίρνοντας πραγματικά πρωτοφανείς διαστάσεις. Ανάλογα ποσοστά πάρα πολύ ψηλά έχει σε, όλα τον, σε όλο τον Ευρωπαϊκό Νότο. Είναι λοιπόν μια μεγάλη πρόκληση για μια χώρα η οποία έχει το ατυχές προνόμιο να είναι η πρώτη στην νεανική ανεργία αυτή την πολύ κρίσιμη στιγμή για την ευρώπη να προχωρήσει πολιτικές και στον τομέα της εκπαίδευσης που να σηματοδοτήσουν μια αλλαγή μια νέα ευκαιρία για τους νέους για μια εκπαίδευση που διατηρώντας τον ουμανιστικό χαρακτήρα της παρόλα αυτά μπορεί να δώσει ένα μήνυμα ελπίδας. είναι πάρα πολύ σημαντικό ειδικά αυτή τη χρονιά των ευρωεκλογών μια χρονιά που κινδυνεύουμε να έχουμε το χειρότερο ευρωκοινοβούλιο που γνώρισε ποτέ η ευρώπη με τον ευρωσκεπτικισμό να ανεβαίνει στα ύψη η νεανική ανεργία θα παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στις επιλογές των πολιτών. ελπίζουμε λοιπόν κύριε υπουργέ από τη θέση σας να μπορέσετε να δώσετε μέσα από τις πολιτικές σας ένα μήνυμα ελπίδας στους νέους της ευρώπης. ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο Υπουργός, μια σύντομη απάντηση δυνατόν. Υπάρχει μια θεματική η οποία διατρέχει οριζόντια και τις τέσσερις ερωτήσεις και της α, κυρίας Μαρή Τερέζ Σάντσε Σμιτ και της κυρίας Παλιαδέλη και του κυρίου Μπόρις και της κυρίας Κοπά. Της κυρίας Κοπά. Αυτή η θεματική, αν με επιτρέπετε να την απαντήσω πρώτα στο βαθμό που μπορώ, αφορά το θέμα της, της ανεργίας, της νεανικής ανεργίας και πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε και βλέπουμε και όλες οι μελέτες μας δείχνουν ότι όλες οι μελέτες του ΩΣΑ αλλά και εθνικές μελέτες μας δείχνουν ότι υπάρχει μια αναντιστοιχία ανάμεσα στις δεξιότητες που χρειάζονται για να μπουν οι νέοι μας και οι νέες μας και να είναι ανταγωνιστικοί στο στίβο της ζωής, στο στίβο της εργασίας και τις δεξιότητες που προσφέρουν, που προσφέρουν τα εκπαιδευτικά μας συστήματα. Αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να σκύψουμε πάνω και να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε και το δεύτερο φυσικά αποτελεί αυτό το οποίο είπατε κυρία Σάντσε Σμί, το θέμα της επαγγελματικής κατάρτισης. Γιατί σε πολλές χώρες, και ιδιαίτερα στη δική μας, αν θέλετε, είναι ένα κλασικό παράδειγμα Ελλάδα, επικράτησε η, η κουλτούρα ότι τα παιδιά μας τα στέλνουμε στο πανεπιστήμιο, γίνονται όλοι γιατροί, δικηγόροι και αυτό απαξίωσε την επαγγελματική εκπαίδευση, την τεχνολογική εκπαίδευση και την κατάρτιση. Αντιστοίχω πρέπει να αναδείξουμε την επαγγελματική τεχνολογική εκπαίδευση και κατάρτιση όχι ω ως ένα αποπέρι τη εκπαίδευση, ω μια δεύτερη διαλογή, ω μια ε, δυνατότητα δεύτερη επιλογής, αλλά ω μια εξίσου σοβαρή επιλογή για τους νέου και τους νέες μα, Για να μπορέσουμε έτσι να έχουμε ένα σωστό εκπαιδευτικό σύστημα κατάρτιση, το οποίο θα δίνει δεξιότητες στου νέου και στι νέες μα και θα τους βγάζει με αξιώσει στην αγορά εργασία αυτό ε, και αναφέρθηκατε στο γερμανικό μοντέλο, το οποίο ε, όσον αφορά το θέμα της μαθητείας, για παράδειγμα, μας δείχνει ένα πολύ, ε, μια σοβαρή επιλογή, όπου μπορούν να συναρθρώσουμε από τη μια το εκπαιδευτικό σύστημα και από την άλλη τους κοινωνικούς εταίρους και τις δυνάμεις της αγοράς. Όλα αυτά λοιπόν, the alliances for apprenticeship, δηλαδή η συμμαχία για τη μαθητεία, είναι μια πολιτική την οποία πρέπει να εφαρμόσουμε. Στην χώρα μου νομοθετήσαμε για πρώτη φορά στην συνολική αναβάθμιση τεχνολογικής εκπαίδευσης και τον τέταρτο χρόνο μαθητείας στα επαγγελματικά και τεχνολογικά λύκεια και έτσι προσπαθούμε να φέρουμε μαζί τις δυνάμεις της αγοράς, μαζί με το εκπαιδευτικό σύστημα και τους νέους ανθρώπους για να αυξήσουμε τις δυνατότητες προσβασιμότητας στην αγορά εργασίας. Αυτή νομίζω είναι μια πολιτική η οποία μπορεί να μας δώσει μια ελπίδα αν την ακολουθήσουμε με σωστά βήματα. Ένα δεύτερο σημείο το οποίο ε, αναφέρατε, κυρία ε, Σάντσε Σμίτ, αφορά φυσικά το θέμα των ε, διαρθρωτικών ταμείων που συμφωνώ απολύτω μαζί σα, όπω και τι δυνατότητε που μα δίνει ο έρασμο, και είναι, είναι ευχής έργων ότι μέσα σε αυτήν την περίοδο τη οικονομικής, βαθιάς οικονομικής χρήσης κατορθώσαμε, κατορθώσατε να πολλαπλασιάσουμε τα, το μπάτζετ, τον προπολογισμό για τον έρασμο που μα δίνει πολύ μεγάλε δυνατότητε. Φυσικά ελπίζω ότι είναι διαδικαστικό το θέμα και ο έρασμος κυρία Παλιαδέλη θα σιγά σιγά θα μεταφραστεί. Είναι, νομίζω ότι θα γίνει αυτό. Συμφωνώ μαζί σας για το θέμα των ανθρωπιστικών επιστημών και αυτό εντάσσεται στη γενικότερη θέαση που πρέπει να έχουμε για την γνώση. Γιατί η γνώση είναι κάτι πολύ ευρύτερο από μια απλή παροχή δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Ουσιαστικά διαμορφώνει χαρακτήρες, και ετοιμάζει τους ανθρώπους για την προσπάθεια της τελείωσης στη ζωή. Είναι κάτι πολύ ευρύτερο. Και πάντοτε το υπόβαθρο θα πρέπει να είναι οι ανθρωπιστικές επιστήμες. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, όλες οι μελέτες μας δείχνουν ότι υπάρχει μια υστέρηση όσον αφορά τις θετικές επιστήμες. Υπάρχει μια υστέρηση στη γνώση μαθηματικών ε, ε, υπολογισμών όσον αφορά τα παιδιά μας και αυτό πρέπει να το δούμε. Και γι' αυτό, και με συγχωρείτε που κάνω πάλι αναφορά για τη χώρα μου, ε, στο νομοσχέδιο για το Λίγιο που ψηφίσαμε ενισχύσαμε τις θετικές επιστήμες γιατί ακριβώς υπήρχε αυτή, αυτή η στέρηση. Αλλά πάντως πρέπει να προσέξουμε και αυτό που μας δείχνουν οι μελέτες και πια και πίζα ότι ε, όσον αφορά την ανάγνωση και εκεί έχουμε μια υστέρηση από, τα, από, τους, ε, από τους νέους μας και αυτό πρέπει εξίσου να, να, προσεχθεί. Περικοπές στην, στον προϋπολογισμό για την εκπαίδευση. Δυστυχώς ζούμε σε μια εποχή που η οικονομική κρίση έχει αγγίξει και τον τομέα της εκπαίδευσης. αλλά είδαμε ότι εάν υπάρξει μια ορθολογική και χρηστή διαχείριση μπορεί να υπάρξει εξοικονόμηση πόρων χωρίς να διακυβεύσουμε την ποιότητα του αγαθού της γνώσης. Εμείς στην, ε, στην Ελλάδα που δυστυχώς πληγήκαμε πολύ από την οικονομική κρίση και δεν ε, ε, ε, κατορθώσαμε να αφήσουμε το εκπαιδευτικό σύστημα εκτός της δημοσιονομικής προσαρμογής, είδαμε ότι με σωστό ορθολογικό σχεδιασμό μπορέσαμε να συμβάλλουμε στη δημοσιονομική προσαρμογή χωρίς να κάνουμε εκπτώσεις στο αγαθό αυτό που λέγεται δημόσια δωρεάν παιδεία και γνώση και παράλληλα κάνοντας σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Θα έλεγα λοιπόν ότι βεβαίως η παιδεία θα πρέπει ε, να έχει πάντοτε έναν αυξημένο προϋπολογισμό, αλλά πάντοτε την ίδια στιγμή θα πρέπει να κοιτάζουμε αυτό να μην σημαίνει κατασπατάληση πόρων. Την ίδια στιγμή να κοιτάζουμε έναν ορθολογικό και χρηστό τρόπο διαχείρισης. Νομίζω ότι αυτά είναι τα πρώτα. Αυτή είναι η πρώτη μου απάντηση. So, uh, ο κύριος Αγκουράκης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, εγώ θα επανέλθω στα ζητήματα που αφορούν τις, ε, την κατάσταση των ε, δαπανών στην παιδεία ε, και γενικά της δημόσιας παιδείας γιατί θεωρώ ότι όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά συνολικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο και όλο και πιο γρήγορα πάμε σε συνθήκες που θυμίζουν μεσαίωνα. Ε, βέβαια όπως ε, ξέρετε κυρία Πρόεδρε από την κρίση δεν υπάρχουν μόνο οι χαμένοι, δεν υπάρχουν μόνο οι άνεργοι και κυρίως οι νέοι άνεργοι. Από την κρίση υπάρχουν και κερδισμένοι. Υπάρχουν πολιεθνικές, υπάρχουν οι πλούσιοι, υπάρχει το μεγάλο κεφάλαιο το οποίο παρά την κρίση και στην Ελλάδα και αλλού γίνεται όλο και πλουσιότερο. Και φυσικά συμβαίνει αυτό γιατί και η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά με την πολιτική της έχω κατά νου Τραπεζική Ένωση, έχω κατά νου Ευρωπαϊκά Εξάμεινα, έχω κατά νου Σύμφωνα Ανάπτυξης και Σταθερότητας, αλλά και μέσω της εκπαίδευσης συμβάλλει, συμβάλλει τα μέγιστα σε αυτή την κατεύθυνση. Είπε ο κύριος υπουργό κάτι που δεν έχει βάση. Ότι δήθεν στην Ελλάδα επειδή οι οικογένειες θέλουν να στέλνουν τα παιδιά τους στα πανεπιστήμια, γι' αυτό έχει απαξιωθεί η επαγγελματική εκπαίδευση. Το ότι στην Ελλάδα κατάφερε η λαϊκή οικογένεια σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ότι πριν τη Χούντα ή στη διάρκεια της Χούντας να στείλει τα παιδιά της στο Πανεπιστήμιο είναι επίτευγμα. Και δεν πρέπει κανείς να την για αυτό το πράγμα. Και μάλιστα σε μια εποχή που μιλάμε για την ανάγκη πολλαπλασιασμού των γνώσεων κτλ. κτλ, κτλ. Αυτό όμως που είναι πραγματικότητα για την επαγγελματική εκπαίδευση και για την ανεργία των νέων είναι κυρίως ότι δεν υπάρχουν δουλειές. Αυτή είναι αλήθεια. Όχι τόσο τα πολλά προβλήματα που έχει το εκπαιδευτικό σύστημα και θα επανέλθω, αλλά κυρίως ότι δεν υπάρχουν δουλειές. Και δεν είναι το θέμα βασικά το ότι δεν είναι προσαρμοσμένο το εκπαιδευτικό σύστημα στις ανάγκες της καπιταλιστικής επιχείρησης, διότι άμα ήταν έτσι, πώς εξηγείται στην Ελλάδα ότι το μεγάλο ποσοστό της ανεργίας είναι νέοι, 60%-62% που υποτίθεται αυτοί οι νέοι είναι πιο κοντά. Έχουν τελειώσει νωρίτερα. Είναι πιο κοντά στι ανάγκε, να το πω έτσι, τη αγορά από ότι είναι οι ηλικιωμένοι. Ποιο, το πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι δεν υπάρχουν δουλειέ και δουλειέ δεν θα υπάρχουν ούτε στο μέλλον. Πολύ περισσότερο που ξέρετε ότι ακόμα και σε συνθήκε όποια ανάκαμψη, όποια και αν εμφανιστεί αυτή, η ανεργία θα είναι ένα μόνιμο και πολύ μεγάλο πρόβλημα και για την Ελλάδα και για άλλες χώρες. Γιατί τέτοια είναι η καπιταλιστική ανάπτυξη σήμερα. Πετάει ζωντανή εργασία. Δεν τους χρειάζεται πια τους εργάτες. Λοιπόν, αλλά επανέρχομαι τώρα στο μοντέλο εκπαίδευσης το οποίο αναπαράγεται και το οποίο παρουσιάζεται. Κύριε Υπουργέ, είναι άραγε τυχαίο που σε δύο σημεία μας είπατε ότι ένα από τα κριτήρια και ένας από τους στόχους της εκπαίδευσης είναι η προετοιμασία των νέων για την επιχειρηματικότητα να τους κάνουμε επιχειρηματίες. Αυτό είναι μια ομολογία για αυτό που είπα, ότι πάμε όλο και περισσότερο στην εποχή του μεσαίων. Διότι οι επιχειρηματίες στην καπιταλιστική κοινωνία που, που ζούμε και δουλεύουν είναι συνώνυμο το εκμεταλλευτή. Θα γίνει μεγάλη πλειοψηφία των νέων, των εργαζομένων επιχειρηματίες και να θέλουν δεν μπορούν. Δεν μπορούν, διότι πάρα πολύ απλά η καπιταλιστική κρίση είναι αυτή που καταστρέφει, κλείνει επιχειρήσεις κτλ. κτλ. Και έχετε το παράδειγμα της Ελλάδα δεν πάω κι αλλού. Αλλά αυτό θέλετε. Αυτό θέλετε και αυτό είναι απόλυτα συμβατό με το χαρακτήρα της κοινωνίας στην οποία ζούμε. Είναι μια καπιταλιστική κοινωνία, είναι μια εκμεταλλευτική κοινωνία και εσείς εργαζόσαστε για να φτιάχνετε το, το πρότυπο του εκμεταλλευτή. Και κλείνω για να εκφράσω πραγματικά την, την αγανάκτησή μας για το γεγονός ότι στην Ελλάδα, όπως ξέρετε πριν μερικές εβδομάδες, έχει ε, ξεκινήσει ένα πρόγραμμα οι δάσκαλοι για την Ευρώπη όπου αναπαράγονται ακόμα και στο δημοτικό αυτές οι απαράδεκτες αξίες της επιχειρηματικότητας, της δίθεν Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες είναι παράγοντας ειρήνης και σταθερότητας αλλά δεν λέτε ότι επί Ευρωπαϊκής Ένωσης έγινε ο πόλεμος στη Ιουγκοσλαβία κτλ. Και τέλος, γιατί και αυτό γίνεται στα ελληνικά σχολεία, το πρόγραμμα ε, «Την Ευρώπη για τους πολίτες» όπου εν καιρό κρίσης μεγάλων ε, ε, ε, λήψεων στην εκπαίδευση ξοδεύονται συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση 228 εκατομμύρια τα επόμενα τέσσερα χρόνια για να εμπεδοθεί ότι ο κομμουνισμός είναι το ίδιο με τον ναζισμό. Γι' αυτό λέω ότι είναι άκρος επικίνδυνη η, η, κατεύθυνση στην εκπαίδευση η οποία υπάρχει σήμερα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε για την ανοχή σας. Ja, Μάλιστα, θα χρειαζόταν μια ολόκληρη μέρα για να τα ανατρέψουμε όλα αυτά. Ε, θα περιορισμούμε, θα περιοριστούμε και στις απαντήσεις κύριε Υπουργέ, φαντάζομαι θα περιοριστείτε σε, στα συγκεκριμένα θέματα. Λοιπόν, για να επανέλθουμε στο θέμα μας κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ πολύ για την ομιλία σας. Διάβασα και τα σχετικά κείμενα που υπάρχουν στο δικτυατικό τόπο μας για την Ελληνική Προεδρία. Ε, είναι πολύ σημαντικά αυτά που θέλετε να κάνετε για την αναβάθμιση της ποιότητας, γιατί όλα αυτά δεν είναι εύκολα εγχειρήματα για σας. Τώρα έχουμε και το νέο ε, πρόγραμμα. Θέλουμε να δούμε και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με το έρασμο Συν. Σας ευχόμεθα κάθε επιτυχία. Λέτε κάπου στα ε, έγγραφά σας ότι θα ε, στηρίξετε το νέο ranking, την ταξινόμηση των πανεπιστημίων. Σε ποια φάση βρίσκεται αυτή η διαδικασία και τι συγκεκριμένα θα κάνετε με το, τη νέα αυτή κατάταξη κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας. Τώρα, στον τομέα της νεολαίας. Θέλετε να προωθήσετε την επιχειρηματικότητα και εδώ δεν θα συμφωνήσω με τον προηγούμενο συνάδελφο. Νομίζω ότι η εκπαίδευση στον τομέα της επιχειρηματικότητας είναι πολύ καλό πράγμα γιατί βοηθάει να, βρεθούν, να βρεθεί απασχόληση, να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας σε πολλούς τομείς. Αυτό είναι θετικό. Ε, και κάτι ακόμα, ίσως ε, είναι μια ευτυχή συγκυρία. Είπατε ότι θα υπάρξουν και δραστηριότητες για τους νέους, θα διοργανώσετε διασκέψεις. Ε, φέτος υποστηρίζεται πολύ η νεολαία η Θεσσαλονίκη, είναι η Ευρωπαϊκή Πόλη των Νέων και χάρη σε αυτή την Επιτροπή. Γιατί η Επιτροπή μας ψήφισε υπέρ και ο συνάδελφος Παπα-Νικολάου ξέρει πολλά για την υπόθεση αυτή. Χαιρόμαστε πάντως που η πόλη αυτή ε, θα είναι ο στόχος των νέων στην Ευρώπη φέτος και έχετε την ευκαιρία να τους δείξετε ότι τους σκέφτεστε, ότι θέλετε να αλλάξετε κάποια αρνητικά. Και κάτι που μου αρέσει επίσης ε, που το έχετε στην ατζέντα σας είναι η προστασία των ε, ανηλίκων και των παιδιών. Είναι πολύ σημαντικό και θα συζητηθεί και αργότερα. Και είναι σημαντικό διότι πολλές φορές ε, ε, κακοποιούνται ε, τα παιδιά στο διαδίκτυο και δεν είναι τόσο στο προσκήνιο αυτό το σοβαρό θέμα όσο θα έπρεπε. Ξέρω ότι για σας είναι προτεραιότητα και πάλι σας εύχομαι κάθε επιτυχία. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, παρατηρώ ότι είναι πραγματικά ένα πρότυπο αυτό που η Ελλάδα, μια χώρα με μεγάλο πολιτισμό, με σπουδαία κληρονομιά, όπως και για την Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι μια ήπειρος που διαθέτει σημαντική κληρονομιά πολιτισμό. Άρα λοιπόν και το μέλλον μας θα πρέπει να είναι συνδεδεμένο με το παρελθόν μας. Βλέπουμε όμως ότι στην Ελλάδα υπάρχει μια βαθιά κρίση. Το ίδιο μπορούμε να μιλήσουμε, το ίδιο μπορούμε να πούμε και για την υπόλοιπη Ευρώπη, ότι αντιμετωπίζει μια βαθιά κρίση. Θα πρέπει λοιπόν να ξεκινήσουμε από τις ρίζες μας από τις ευρωπαϊκές μας ρίζες, από τις ευρωπαϊκές μας αξίες, από το ευρωπαϊκό μας παρελθόν και να το προσαρμόσουμε, να προσαρμόσουμε την κληρονομιά μας στο μέλλον μας. Αυτό που εύχομαι είναι η ελληνική προεδρία να καταφέρει να ακολουθήσει αυτό το πρότυπο και να αποτελέσει ένα παράδειγμα. Να μπορέσει να προετοιμάσει αυτό το μελλοντικό πρότυπο για την Ευρώπη. Και όσον αφορά τα πανεπιστήμια, υπάρχουν στατιστικές. Σύμφωνα με τις στατιστικές αυτές, ανάμεσα στους νέους υπάρχουν πάρα πολλοί που διαθέτουν διπλώματα, αλλά Ακριβώς όσο περισσότεροι νέοι έχουν σπουδάσει, τόσο χαμηλότερο είναι το ποσοστό ανεργίας. Η εκπαίδευση, η παιδεία, οι σπουδές βοηθούν να επιβιώσει κανείς σε αυτή την περίοδο κρίσης. Αυτό ισχύει και για τη Ρουμανία και για άλλες πρώην κομμουνιστικές χώρες. Και θα πρέπει ακριβώς να προσέξουμε την εκπαίδευση, την παιδεία. Είναι πολύ σημαντική τομή. Δεν μπορούμε να μείνουμε πίσω, να αργοπορήσουμε, να βραδιπορήσουμε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και να το πετύχουμε και στις χώρες ε, που, στις οποίες αναφέρθηκα προηγουμένως. Και θα πρέπει να ακολουθήσουμε το δρόμο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Εμφανίζονται όμως και προβλήματα και στα οποία δεν είμαστε σύμφωνοι όσον αφορά τους τρόπους επίλυσης. Ε, μιλάνε πολύ για την κινητικότητα, αλλά είναι καρνητικό αυτό. Την Ουγγαρία, τη Ρουμανία, την Τρασιλβανία, τόσες πολλές χώρες εγκαταλείπονται από την νεολαία και η χώρα παραμένει στα αυτά τα επίπεδα τα παλιά γιατί ο νέος αυτός κόσμος που φεύγει δεν επιστρέφει για να μας βοηθήσει να επιστραφεί η γνώση που έχει αποκτηθεί στις δυτικές χώρες. Τη χρειαζόμαστε στις χώρες μας εμείς αυτή τη γνώση για να αποτελέσουμε μέρος του ανεπτυγμένου κόσμου. Άρα λοιπόν, όχι μόνο υπέρ της κινητικότητας, θα πρέπει να παροτρύνουμε τους νόους, τους νέους να παραμείνουν στη χώρα, να βρουν μια δουλειά, να παραμείνουν στη χώρα τους γιατί θα πρέπει ανάμεσα στην ανατολική πλευρά της Ευρώπης, η δυτική, να υπάρξει μια ισορροπία. Και μετά όταν μιλάμε για τις αξίες της Ευρώπης, μιλάμε και για την αξία των εργατικών χεριών σαν εμπόρευμα. Είναι όμως σημαντικότατες και οι ηθικές αξίες. οι αξίες που εκφράζει η Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι χώρα χριστιανική και αντιπροσωπεύει τις χριστιανικές μας ρίζες. Παρά, συνδυσμένο παράδειγμα είναι εντάξει η αξία της εργασίας. Οι Βέλγοι, οι Βρετανοί, οι Γάλλοι, δεν θέλουν να δεχτούν ε, να κάνουν ορισμένε εργασίες ε, γιατί τις θεωρούν ε, βρώμικες εισαγωγικά δουλειές είτε χειρονακτικές. Χρειάζεται λοιπόν την εισαγωγή εργατικών χεριών αλλά θα πρέπει να προσέξουμε και την ηθική αξία της εργασίας. Θα πρέπει να τη διδάξουμε στους νέους, να την μάθουν οι νέοι. Γιατί δεν είναι ότι αυτόματα γίνεται κανείς ευτυχισμένος αν γίνει επιχειρηματίας. Υπάρχει η αγάπη με την ευρύτερη της έννοια σαν αξία. το Ευαγγέλιο να ξαναισχύσει στην Ευρώπη, οι αξίες του. Μια Ευρώπη λοιπόν που να βασίζεται και σε αυτές τις αξίες. Θέλουμε την αναγέννηση μιας παρόμοιας Ευρώπης. Ευχαριστώ κύριε Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, θα μιλήσω ελληνικά για να τιμήσω την Προεδρία. Κύριε Υπουργέ, καλώ ήρθατε. Εύχομαι καλή δύναμη και καλή επιτυχία στην ελληνική Προεδρία, μια Προεδρία που διεξάγεται σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο και δύο ερωτήσεις, πολύ σύντομα. Το πρώτο σχόλιο είναι ότι σε αυτήν την επιτροπή τα χρόνια που πέρασαν, αναφέρθηκε η κυρία Νεβεντάλοβα, σε διάφορα θέματα δουλέψαμε σε βάθος. Και τα κείμενα που ψηφίστηκαν ως αποτέλεσμα της συζήτησης και της διαβούλευσης ε, ε, ε, περιέχουν πολλά μηνύματα τα οποία σε πολλές περιπτώσεις είναι καινοτόμα, αποτελούν κατευθύνσεις που αν υιοθετηθούν μπορούν να οδηγήσουν και σε λύσεις. Επειδή ξέρετε υπάρχει το ζήτημα τη συμπληρωματική αρμοδιότητα, επικουρικότητα, αισθανόμαστε κάποιε φορέ ότι αυτά που ψηφίζουμε δεν ακούγονται όσο δυνατά θα θέλαμε στα κράτη-μέλη και δεν υιοθετούνται. Ε, άρα η πρώτη παράκληση είναι αυτή, επειδή είμαστε και πριν από τι εκλογέ, η Ελληνική Προεδρία να αναδείξει τα μηνύματα αυτή τη Επιτροπή. Ε, θα ήθελα να κάνω δύο σύντομα ερωτήματα, επειδή ε, δούλεψα και εγώ πολύ σε ό,τι αφορά τη στρατηγική για την νεολαία. Το, το πρώτο ερώτημα είναι ε, πώς σκέπτεστε να προωθήσετε και εσείς και να αναδείξετε και να αναλύσετε το ζήτημα των ανοιχτών δομών εκπαίδευσης όπως προκύπτουν σήμερα και με τις νέες τεχνολογίες, τα open educational, τα, open resources που κουβεντιάσαμε και σήμερα το πρωί στην Επιτροπή μας, τι σκοπεύετε, που είναι πολύ σημαντικό δεδομένο πλέον και για τα νέα παιδιά σε όλη την Ευρώπη, πώς σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε το ζήτημα της άδεια χρήσης, τα copyrights, όλα αυτά τα θέματα. Η δεύτερη ερώτηση αφορά, επειδή εντάξει, δεν θα ήθελα και εγώ να, να αναφερθώ όπω έκανε ο εκλεκτό συνάδελφο ο κ. Αγκουράκη προηγουμένω σε εθνικά ζητήματα, αλλά εν πάση περιπτώσει επειδή είμαστε μέσα στην κρίση, πώ σκοπεύετε να ενισχύσετε ω Προεδρία, και αυτό βεβαίω αφορά και την Ελλάδα, το, το ζήτημα τη σύνδεση εκπαίδευση με την αγορά εργασία ακόμη πιο στενά. Θυμάστε πριν από ένα-ενάμιση χρόνο περίπου, μαζί και με την Πρόεδρο τη Επιτροπή μα, είμαστε σε μια εκδήλωση και κουβεντιάζαμε για το λεγόμενο dual system που έχει και η Γερμανία το αναφέρατε και πριν και πώς σκοπεύετε και με την μεταρρύθμιση που κάνετε στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα να το κάνετε αυτό ε, και να το μεταδώσετε ως μήνυμα και σε όλη την Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Thank you. We have noch Η κυρία Τρούπαλ. Δύο ομιλητές έχουμε ακόμα. Ευχαριστώ Υπουργέ για την ομιλία σας. Μία συγκεκριμένη ερώτηση θα κάνω μόνο. Μιλήσατε για τα ανοιχτά διαδικτυακά ή επιγραμμικά μαθήματα. Τα MOOCs. Ποια κάλυψη ε, επιτυγχάνουν στα ελληνικά πανεπιστήμια και σχολεία για να έχουμε έτσι μια ιδέα για ποιο πράγμα, για ποια τάξη μεγέθους μιλάμε. Πολύ ωραία. Σύντομα και σαφή αυτά που είπατε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Να ευχηθώ ότι καλύτερο στην Ελλάδα και σε εσά, κύριε Υπουργέ. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία στην Προεδρία σας. Θα είμαι και εγώ συντομότατος με μια σύντομη ερώτηση. Καταρχήν να ζητήσω συγγνώμη που καθυστέρησα γιατί έπρεπε να παρευρεθώ και σε μια άλλη συνεδρίαση. Εμείς εγκρίναμε τον προϋπολογισμό, εγκρίναμε προγράμματα, ε, έργα, είμαστε στην αρχή του νέου δημοσιονομικού πλαισίου. Ερωτώ λοιπόν, οι πολίτες μας περιμένουν να δουν να αρχίσουν καινούργια προγράμματα, έργα ε, που θα χρηματοδοτηθούν με ευρωπαϊκά κονδύλια. Υπάρχει χρονοδιάγραμμα τώρα για τα ευρωπαϊκά αυτά κονδύλια. Δηλαδή μπορούν να ξεκινήσουν τα προγράμματα γιατί μας ρωτούν οι πολίτες της Ευρώπης, των χωρών μας, τι, τι γίνεται. Τα χρήματα για το 2014 θα εξαρτηθούν από την υπογραφή της Συμφωνίας Σύμπραξης ή Εταιρικής Σχέσης με τα κράτη-μέλη. Εξαρτώνται και από την έγκριση των ε, ε, ε, επιχειρησιακών προγραμμάτων. Τι απαιτείται. Μπορούμε να αρχίσουμε δηλαδή να ε, μοιράζουμε τις αιτήσει για να τις συμπληρώσουν ή όχι τώρα τον Ιανουάριο του 2014 γιατί μιλάμε για προγράμματα ανταλλαγών φοιτητών και με ρωτούν απευθείας πότε μπορούμε να υποβάλουμε την αίτηση, πότε θα πρέπει να αρχίσουμε με τις αιτήσει. Ευχαριστώ και καλή επιτυχία. Mr. Minister, please. Υπουργέ. Thank you. Να αρχίζω ε, δίνοντας μια, προσπαθώντας να δώσω μια απάντηση στα όσα είπε ο κύριος Σαγκουράκης όσον αφορά τα θέματα α, της εκπαίδευσης, της εισαγωγής στα πανεπιστήμια και της επαγγελματικής τεχνολογικής εκπαίδευσης. Προφανώς είναι επίτευγμα αυτό το οποίο έγινε όσον αφορά την προσβασιμότητα στα τριτοβάθμια, α, τα εγκεντρήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Δεν μιλώ γι' αυτό. Λέγω κάτι άλλο, ότι οδηγηθήκαμε σε μια στρέβλωση γιατί δώσαμε μεγάλη έμφαση παραγνωρίζοντας τις δυνατότητες αλλά και την ε, ε, αξία της επαγγελματικής και τεχνολογικής εκπαίδευσης. Αυτό στην, χώρα μας, αλλά αυτό έγινε και σε άλλες χώρες. Αυτό είχε, μια, είχε ένα αποτέλεσμα, είχε ως αποτέλεσμα την απίσχναση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων της κοινωνίας μας, των νέων μας και του εργατικού μας του εργατικού δυναμικού. Αυτό επίσης είχε ένα αποτέλεσμα στην, στον παραγωγικό ιστό όσον αφορά την, ε, την ε, οικονομική δυσπραγία και την απίσχναση του παραγωγικού ιστού ιδίως στη χώρα μας. Αυτό που λέμε λοιπόν είναι ότι η επαγγελματική εκπαίδευση δεν πρέπει να είναι μια δυνατότητα δευτέρας διαλογής, μια επιλογή δεύτερης διαλογής. Πρέπει να είναι εξίσου σημαντικό να είναι κάποιος δικηγόρος, γιατρός, με το να είναι τεχνίτης, δεξιοτέχνης, τεχνολόγος. Είναι θέμα επιλογής και αυτό πρέπει να δίνουμε την δυνατότητα ίδιας ποιότητας εκπαίδευσης. Τώρα, όσον αφορά για το θέμα της προετοιμασίας για την επιχειρηματικότητα σε ένα καπιταλιστικό μοντέλο ανάπτυξης, προφανώς ε, είπα πρώτος ότι η, η γνώση και η παιδεία είναι πολύ περισσότερα από την στενή σχέση με τον ε, τρόπο των παραγωγής και την αγορά, αλλά δεν μπορεί να είναι αποκομμένη η διαδικασία απόκτησης γνώση από την αγορά και από την ε, επιχειρηματικότητα και από την οικονομία. Τώρα, το καπιταλιστικό μοντέλο ανάπτυξης, εξ όσο γνωρίζω, είναι το μόνο μοντέλο που υπάρχει στην οικονομία στον κόσμο, άρα νομίζω ότι γι αυτό, αυτό υπάρχει και γι' αυτό προετοιμάζουμε του νέου και τι νέε μα όσον αφορά το θέμα της προετοιμασίας και της δασκαλίας στα σχολεία μας για την Ευρώπη και τους πολίτες είναι ένα πρόγραμμα για το οποίο είμαστε υπερήφανοι γιατί πέρα από την εθνική συνείδηση νομίζω ότι πρέπει να εδρεωθεί και η ευρωπαϊκή συνείδηση ότι είμαστε πολίτες της Ευρώπης. Αυτό το οποίο είπε η κυρία Νεβεντάλοβα όσον αφορά το, θέμα του το, Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική πρωτοβουλία γιατί μας δίνει μια συγκεκριμένη ευρωπαϊκή μορφή κατάταξης, γιατί συγκρίνει τα ιδρύματα, τα ανώτατα εκπαιδευτικά μας ιδρύματα, όχι μόνο στον τομέα της έρευνας αλλά και της διδασκαλίας. Είναι σημαντικό. Έχουμε την πρώτη συλλογή δεδομένων πραγματοποιήθηκε νομίζω τον Δεκέμβριο του του 2013 και η πρώτη κατάταξη πρόκειται να δημοσιευτεί και νομίζω ότι πολλά ιδρύματα πέρα από 400-500 ήδη έχουν συμπεριληφθεί σε αυτόν τον κατάλογο και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα μας απασχολήσει και θα διοργανώσουμε ένα συνέδριο για να δούμε τα πρώτα αποτελέσματα. Όπως επίσης σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αυτό το οποίο μας απασχολεί είναι το θέμα των συγχωνεύσεων των πανεπιστημίων και των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Και είναι μια διαδικασία η οποία μας μας απασχόλησε στην Ελλάδα με το σχέδιο Αθηνά. Συγχωνεύσαμε 104 τμήματα και 4 ιδρύματα, αλλά βλέπουμε ότι είναι μια ευρωπαϊκή διαδικασία, τη βλέπουμε ότι μελετάται και στη Γαλλία και σε άλλες χώρες και νομίζω ότι είναι μια διαδικασία που δεν υπόκειται μόνο σε όρους δημοσιονομικής προσαρμογής ή δεν ανταποκρίνεται μόνο στην οικονομική κρίση, αλλά ανταποκρίνεται και σε συνέργειες δυνάμεων, σε δημιουργία ισχυρότερων οργανισμών, πιο ανταγωνιστικών, οι οποίοι με εξωστρέφεια και με βάση την αριστεία μπορούν να είναι ανταγωνιστικοί σε διεθνές επίπεδο. Συνεπώς και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο μας απασχολεί, όπως αυτό το οποίο θέσατε και είναι πάρα πολύ σημαντικό, για το ζήτημα της κακοποίησης των παιδιών, το οποίο θα το ενέτασα, αν θέλετε, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο που έχει να κάνει με τα ανθρώπινα δικαιώματα των παιδιών. Και γιατί παρατηρούμε ότι ένα, πολύ, ένα από τα ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε είναι το περίφημο bullying στα σχολεία και είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει όλους, μας απασχολεί ιδιαίτερα και μας ως χώρα αλλά και νομίζω και ε, γενικότερα τον, ε, την Ευρώπη Υπάρχουν πάρα πολλές πρωτοβουλίες πάνω σε αυτό το επίπεδο και νομίζω ότι πρέπει μια και καλή να ξεριζώσουμε αυτό το φαινόμενο μέσα από τα εκπαιδευτικά μας συστήματα, να φέρουμε την ανοχή στη διαφορετικότητα, να φέρουμε την, την, την εκμάθηση της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών, γιατί αυτό ουσιαστικά μορφώνει πολίτες οι οποίοι αύριο από θέση ευθύνης θα μπορέσουν να ξεριζώσουν και την κατάρα του πολέμου μια και καλή από, το, από, το, από, τον κόσμο. Συνεπώς αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα το οποίο μας απασχολεί πάρα πολύ. Και όσον αφορά το θέμα της, που έθεσε ο κύριος Λάσλο Τόρες, όσον αφορά το θέμα της κινητικότητας, προφανώς η κινητικότητα είναι πια μια πραγματικότητα μέσα σε ένα παγκοσμιοποιημένο χώρο η κινητικότητα σε μια ε, παγκοσμιότητα, η κινητικότητα είναι εκ των όνου κάνευ και δεν είναι μόνο κινητικότητα για τη μάθηση, είναι κινητικότητα κεφαλαίου, κινητικότητα ανθρώπων, κινητικότητα εμπορευμάτων. Υπάρχει αυτό, είναι μια πραγματικότητα, δεν μπορούμε να την αγνοήσουμε και άρα πρέπει να το δούμε πώς αυτό μας, ε, και στη μάθηση μας δίνει συγκριτικά πλεονεκτήματα. Και φυσικά βέβαια πάντοτε μιλάμε α, και καλά κάνετε και το υπενθυμίζετε για μια ε, εκπαίδευση για ένα εκπαιδευτικό σύστημα το υπόβαθρο του οποίου βέβαια θα έχει ένα αξιακό σύστημα. Δεν μπορούμε να μιλάμε για μια ε, παιδεία δυνατοτήτων χωρίς να υπάρχει στο υπόβαθρο ένα αξιακό σύστημα. Ο, ο κύριος Παπα-Νικολάου έθεσε τα θέματα ε, της σύνδεσης της αγοράς με την εκπαιδευτική διαδικασία. Όπως ε, αναφέραμε υπάρχει το διτό σύστημα, το dual track system, το οποίο είναι ένα, μια πολύ σοβαρή προοπτική την οποία εμείς υιοθετήσαμε στην Ελλάδα μετά από πολλά χρόνια εφαρμόσαμε το τέταρτο χρόνο μαθητείας και αυτή τη χρονιά φέρνουμε ε, κοντά χωρίς να περιμένουμε να φτάσουμε, γιατί τώρα νομοθετήσαμε το, το νέο επαγγελματικό λύκειο, χωρίς να περιμένουμε να φτάσουμε τον τέταρτο χρόνο για να υιοθετήσουμε τη μαθητεία, κάνουμε μια πρόσκληση ώστε οι απόφοιτοι από τα επαγγελματικά τεχνολογικά λύκεια της τελευταίας εξαετίας να έρθουν σε ε, συνάφεια με τους κοινωνικούς εταίρους, με την αγορά, με επιχειρήσεις, για να μπορέσουμε να έχουμε ένα χρόνο μαθητείας. Αυτό μας, δίνει, ε, μας δημιουργεί λοιπόν μια κουλτούρα όπου και οι επιχειρήσεις και η αγορά και οι κοινωνικοί εταίροι επενδύουν στους, ε, στους μαθητές μας, στους αυριανούς εργαζόμενους με μια πιο μακρόχρονη σχέση η οποία δεν έχει τα χαρακτηριστικά αυτό που λέγαμε internship, έτσι, που ήταν κάτι εντελώ επιφανειακό και, όχι μεθοδευμένο. Συνεπώς αυτό είναι μια πολιτική η οποία προσδοκούμε ότι θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο και οι δύο πλευρές βλέπουν ε, τα πράγματα, θα φέρει κοντά εκπαιδευτικό σύστημα και αγορά και νομίζω ότι τα αποτελέσματα θα είναι θετικά για, την, ε, για τους νέους και τις νέες μας. όσον αφορά το ζήτημα των ε, online courses τα, που έθεσε η κυρία Τρόπελ. Εδώ έχουμε, ε, είμαστε στην, ε, σε μια περίοδο που αυτό διαδίδεται, αν θέλετε, ε, στον χώρο μας. Έχουμε το, εθνικό, έχουμε το ανοιχτό πανεπιστήμιο, το οποίο α, ακριβώς είναι μάθηση εξ και σιγά σιγά φέρνουμε αυτήν την δυνατότητα των online courses αλλά όπως είπαμε αυτό πρέπει να δει και πρέπει με πολύ μεγάλη σοβαρότητα να αντιμετωπίσουμε και προβλήματα τα οποία αναφύονται μέσα από αυτό που έχουν να κάνουν με, το, τα ζητήματα των πνευματικών δικαιωμάτων, με το ποιο διδάσκει την πιστοποίηση, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία πρέπει να, να τα δούμε συνολικά. Και επίσης αυτό το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα με, με προγράμματα να ε, ε, εδραιώσουμε κυρίως ε, στη δική μας περίπτωση είναι το ψηφιακό σχολείο, δηλαδή η δυνατότητα πρόσβασης σε αυτή την τεχνολογία που θα μπορέσουν ε, ακόμα και σε, με τις ιδιαιτερότητες που εμείς αντιμετωπίζουμε με απομακρυσμένα σχολεία σε νησιωτικές στις ορεινές περιοχές να μπορέσουμε να έχουμε μια δυνατότητα σε τέτοιες τεχνολογίες που θα μας αυξήσουν τις μαθησιακές δυνατότητες. Τώρα, για τα έργα που χρηματοδοτούνται, νομίζω αμέσως πρέπει να γίνουν επίσης, γιατί αυτό ε, εντάσσεται μέσα στο 2014. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Χθες και σήμερα μιλήσαμε για αυτούς τους ανοιχτούς πόρους, ανοιχτούς εκπαιδευτικούς πόρους. Πιστεύουμε ότι υπάρχουν και γεωγραφικά εμπόδια τα οποία τώρα θα τα ξεπεράσουμε με τους ανοιχτούς εκπαιδευτικούς πόρους. Σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας. Απαντήσατε σε όλες τις ερωτήσεις και τις συμπληρωματικές. Υπογραμμίζω και εγώ αυτό που είπατε. Αγαπητέ συνάδελφε Αγκουράκη, είπατε ότι είπε ο Υπουργός ότι θέλουν τους νέους να τους κάνουν επιχειρηματίες. Μα χωρίς επιχειρήσεις δεν θα υπάρχουν θέσεις εργασίας. Αυτό πρέπει ο καθένας να το ξέρει. Δεν δημιουργούνται από το κράτο και τη διοίκηση θέσει εργασία, αλλά από του επιχειρηματίε. Γι' αυτό χρειαζόμαστε καλά εκπαιδευμένου επιχειρηματίε που θα δίνουν στον κόσμο εργασία. Παντού ισχύει αυτό σε κάθε κράτο και δεν έχει να κάνει με τον καπιταλισμό. Πρόκειται για την ε, απλή πραγματικότητα. Άρα νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο, θα τον ακολουθήσαμε από κοινού και είπατε ότι το θέμα δεν είναι μόνο να έχουμε τριτοβάθμια εκπαίδευση, ανώτατη εκπαίδευση, αλλά εκπαίδευση, παιδεία, γιατί χρειαζόμαστε μορφωμένους ανθρώπους και τεχνικώς καταρτισμένους και ξυλουργούς και υδραυλικούς, ε, τεχνικούς τεχνίτες όλων των ειδών. Αυτά είναι επαγγέλματα πολύ σημαντικά για την καθημερινότητά μας. Όμως θα πρέπει και η κοινωνία να το καταλάβει και να αποδεχθεί αυτά τα επαγγέλματα και να τα εκτιμήσει όπως τους αξίζουν. Εκεί πρέπει να δουλέψουμε. Όμως ε, δεν μπορεί να γίνει αυτό μόνο με υπαγορεύσεις και νόμους. Θα πρέπει μέσα στην κοινωνία να τα καταφέρουμε. Κάτι ακόμα που νομίζω ότι πρέπει να το αναδείξουμε. Ε, όπως το Κομένιους, το παλιό πρόγραμμα του Έρασμος ΣΥΝ, ε, έχουμε τη δυνατότητα περισσότερο την ε, εκπαίδευση και την κατάρτιση να την προωθήσουμε περισσότερο για τους εκπαιδευτικούς. Αυτό το πορόβλεψε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλοι είμαστε σε καλό δρόμο. Διότι αν επενδύσουμε μαζικά εκεί θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Όχι μόνο στους ανοιχτούς εκπαιδευτικούς πόρους αλλά και σε πολλούς άλλους τομείς. Και πάλι σας ευχαριστώ πολύ. Ε, δεν ξέρω αν η Κομισιόν θέλει να μας απαντήσει σε αυτό το σημείο σε κάποιες ερωτήσεις που έγιναν. Μου φαίνεται μιλάνε μεταξύ τους, ας τα να το κάνουμε την άλλη φορά. Ε, όχι, όχι θέλει να μιλήσει. Α, ναι, στα γρήγορα να μας πείτε πότε θα μεταφραστούν τα κείμενα. Τα κείμενα του έρασμου συν πότε θα μεταφραστούν σε όλες τις επίσημες γλώσσες, για παράδειγμα. Και ο κύριος Μάτουλα έκανε την ερώτηση πότε θα αρχίσουν οι εργασίες για όλα αυτά τα προγράμματα. Γιατί εγώ έχω την εντύπωση βέβαια ότι έχουμε αρχίσει εδώ και καιρό να δουλεύουμε πάνω σε αυτά, αλλά να του το πείτε και εσείς ο ίδιος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να σας το αποσαφηνίσω. Το κείμενο έχει μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες και η πρώτη πρόσκληση προσφορών κατά τα Χριστούγεννα, πρέπει να το ξέρει ο κύριος Μάτιλα, έχει αρχίσει 12 Δεκεμβρίου πριν τα Χριστούγεννα και αυτή έγινε σε όλες τις γλώσσες αλλά το κείμενο είναι μακροσκελές, υπάρχει ένα μακροσκελές πρόγραμμα που δεν έχει ακόμα μεταφραστεί, είναι ο, το λεπτομερές πρόγραμμα και ο οδηγός κυρίως χρήσης του προγράμματος. Αυτό είναι 300 σελίδες περίπου, δεν έχουν ακόμα μεταφραστεί όλες. Αλλά τους επόμενους μήνες θα υπάρξει και αυτό μεταφρασμένο. Και προς την κυρία Παλιαδέλη θα μπορούσα να πω ότι αν κανείς έχει μια δυσκολία για πρόσβαση για τον οδηγό αυτό στα ελληνικά, τότε μπορεί να απευθυνθεί σε ελληνικές αρχές που είναι έτοιμες να του δώσουν οδηγίες ως προς το πώς να έχει πρόσβαση στον οδηγό στο πρόγραμμα. Πάντως υπάρχει, όχι δεν είναι αυτό το πρόβλημα της Ελλάδας ή όχι, μου έχουν πει ότι δεν έχει μεταφραστεί σε καμία άλλη γλώσσα εκτός από τα αγγλικά. Ισχύει αυτό. Εμείς ξέρουμε ελληνικά και αγγλικά, δεν είναι το πρόβλημα της Ελλάδας. Καλώς νεύεται καταφατικά, ακόμα δεν έχει μεταφραστεί σε άλλη γλώσσα, μόνο στα αγγλικά υπάρχει και σας λέω ότι αυτό δεν αρκεί. Πρέπει να γίνουν οι μεταφράσεις. Το χρόνο τον είχατε, αξιοποιήστε το, μη μας λέτε τους επόμενους μήνες, σε τέσσερι εβδομάδε να τελειώσουν. Υπάρχουν παντού καλοί μεταφραστές, έχουμε και εδώ και αλλού και εσεί το δικό σα οίκο. Λοιπόν, κοιτάξτε το αυτό, είναι σημαντικό γιατί χρειάζεται η μετάφραση για κάποιον που θέλει να το χρησιμοποιήσει. Αυτό είναι μια φιλική υπόδειξη προς την Κομισιόν. Παρακαλώ, ανταποκριθείτε σε αυτήν, ακολουθήστε την. Η κυρία Παλιαδέλη σωστά τα είπε. Ε, οι προκηρύξεις όμως υπάρχουν σε κάθε γλώσσα. Έτσι υπάρχει, αν, σας κατάλαβα καλά, ε, υπάρχουν στην κάθε γλώσσα. Ευχαριστώ και πάλι Υπουργέ. Κάθε επιτυχία να εκπληρωθούν όλες ε, οι επιθυμίες που εκφράσαμε και παρακαλώ τώρα να έρθει ο επόμενος Υπουργός. για τις ερωτήσεις. Και αν ε, όποτε κρίνει το Κοινοβούλιο ότι υπάρχουν θέματα για ερώτηση, εγώ είμαι στη διάθεση να έρθω να απαντήσω. Yeah, okay. Thank you. Ωραία, ευχαριστούμε. So. Uh, Ο κύριος Παναγιωτόπουλος είναι μαζί μας τώρα, Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού. Έχουμε πολλές ε, ερωτήσεις που δεν απαντήθηκαν και νομίζω ότι είναι κατάλληλη στιγμή να μιλήσουμε με τον ε, Υπουργό Πολιτισμού και Προεδρεύοντα του Συμβουλίου. Ε, είχαμε μετά το 2020 μια Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Πολιτισμού και θα ακούσαμε και για την έκθεση της Βερζιά που ψηφίστηκε σήμερα, την οδηγία για την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών που παρανόμως απομακρύνθηκαν από μια χώρα μέλος είναι κατάλληλη στιγμή αυτή επί ελληνικής προεδρίας να το συζητήσουμε. Έχουμε λοιπόν ε, τα θέματα αυτά που ε, εσείς μπορείτε να ολοκληρώσετε επί της Προεδρίας σας. Τα πολιτιστικά θέματα που μπορείτε να τα λύσετε, ε, έχουμε εμπιστοσύνη ότι θα τα λύσετε. Έχουμε εμπιστοσύνη ε, στην ε, κατανόησή σας σχετικά με τα οράματα αυτού του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, εξοχότατα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Για μένα είναι μεγάλη τιμή και ευχαρίστηση η παρουσία μου εδώ στις Βρυξέλλες και η ευκαιρία που μου δίνεται να σας παρουσιάσω τις προτεραιότητες της ελληνικής προεδρίας ιδιαίτερα για θέματα αθλητισμού και πολιτιστικών. Θα ήθελα να σας συγχαρώ, κυρία Πρόεδρε, καθώς και όλα τα μέλη της Επιτροπής σας, γιατί τον Μάιο θα οργανωθούν οι ευρωπαϊκές εκλογές. Να σας ευχαριστήσω λοιπόν για τις προσπάθειες και τα επιτεύγματά σας κατά την θητεία αυτή. Τώρα, για τις προτεραιότητες της ελληνικής προεδρίας επιτρέψτε μου να συνεχίσω στην μητρική μου γλώσσα. Κυρίες και κύριοι μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο πολιτισμός αποτελεί έναν τομέα στρατηγικού ενδιαφέροντος για την Ελλάδα, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί και έναν τομέα στρατηγικού ενδιαφέροντος για ολόκληρη την Ευρώπη. Ο πολιτισμός παίζει καθοριστικό ρόλο για τις σχέσεις της σύγχρονης Ευρώπης με τον υπόλοιπο κόσμο. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να συζητήσουμε και στην Ευρώπη για μια κοινή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα θέματα του πολιτισμού που θα αφομοιώνει δημιουργικά την ιστορία τις γλώσσες και τις παραδόσεις των λαών που απαρτίζουν σήμερα το ευρωπαϊκό οικοδόμημα και συναποτελούν τον κοινό μας ευρωπαϊκό πολιτισμό. Ο πολιτισμός όλες τις εκφάνσεις του αποτελεί ένα από τα, από τα μεγάλα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ευρώπης. Ιδίως σε μια εποχή όπου επικρατούν δυσμενείς οικονομικές συνθήκες και κοινωνικές ανισότητες ο πολιτισμός μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά και στην οικονομική ανάκαμψη και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής ως καθοριστικός παράγοντας στη διαμόρφωση ταυτότητας και ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης. Στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020 αλλά και σε σχέση με το ρόλο του πολιτισμού ως πυλών ανάπτυξης η ελληνική προεδρία θα συνεισφέρει σημαντικά στη συζήτηση για το ρόλο τον οποίο καλούνται να διαδραματίσουν η πολιτιστική κληρονομιά και η δημιουργική οικονομία τον 21ο αιώνα. Για τα θέματα αυτά η Ελληνική Προεδρία θα πραγματοποιήσει δύο συνέδρια. Θα εκπονηθούν δε συμπεράσματα από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Η συμβολή του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα και ιδιαίτερα της πολιτιστικής κληρονομιάς στη βιώσιμη ανάπτυξη». Ειδικότερα, η Ελληνική Προεδρία θα εστιάσει την προσοχή της στην οικονομική και κοινωνική διάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς διερευνώντας ταυτόχρονα θεματικές όπως οι καινοτόμοι τρόποι χρηματοδότησης οι οικονομικές και κοινωνικές συμπράξεις η διεύρυνση του ακροατηρίου και η κοινωνική συνοχή. Έμφαση επίσης θα δοθεί στην ανάγκη διαμόρφωσης και προώθησης μιας κοινή ευρωπαϊκής προσέγγισης για την πολιτιστική κληρονομιά στο πλαίσιο αυτής της προτεραιότητας οργανώνουμε συνέδριο με τίτλο «Η πολιτιστική κληρονομιά στο προσκήνιο προς μια κοινή προσέγγιση για μια βιώσιμη Ευρώπη» από τις 6 ως τις 8 Μαρτίου στο νέο Μουσείο της Ακρόπολης στην Αθήνα. Επιπλέον η Προεδρία θα αναδείξει θέματα σχετικά με την αυξανόμενη σπουδαιότητα του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα θα εξεταστούν παράμετροι όπως η πληροφόρηση για τα υπάρχοντα εργαλεία και την τεχνογνωσία που διευκολύνουν την πρόσβαση στη χρηματοδότηση οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της καινοτομίας με γνώμονα και κριτήριο την επιχειρηματικότητα αλλά και οι αποτελεσματικές στρατηγικές για την κοινωνική και οικονομική ευημερία. Για το θέμα αυτό η Ελληνική Προεδρία οργανώνει ένα άλλο συνέδριο με τίτλο Χρηματοδοτώντα τη δημιουργικότητα» 20 και 21 Φεβρουαρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Κυρίες και κύριοι, η Ελληνική Προεδρία επιθυμεί να συνεχιστεί ο διάλογος για τον σημαίνοντα ρόλο του πολιτισμού στις εξωτερικές, στις διεθνείς σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις διεθνείς διαδικασίες λήψεως αποφάσεων. Για το σκοπό αυτό διοργανώνουμε στην Αθήνα στις 17 Ιουνίου άτυπη συνάντηση υψηλών αξιωματούχων των Υπουργείων Πολιτισμού και Εξωτερικών αρμοδίων για τις εξωτερικές πολιτιστικές σχέσεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το συνέδριο θα γίνει στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Στη συνάντηση θα δοθεί έμφαση στον διαπολιτισμικό διάλογο, τις αμοιβαίες πολιτιστικές ανταλλαγές και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας. Σε σχέση με το πρόγραμμα εργασίας 2011-2014 για τον πολιτισμό, η Ελληνική Προεδρία έχει σκοπό να ενθαρρύνει το διάλογο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του όπως επίσης και την προετοιμασία των θεματικών προτεραιοτήτων για το νέο πρόγραμμα. η προεδρία θα αναλάβει επίσης τις διαπραγματεύσεις με το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ώστε να επιτευχθεί συμφωνία για την αναδιατύπωση της οδηγίας 93 7 του Συμβουλίου σχετικά με την επιστροφή των παρανόμως εξαχθέντων πολιτιστικών αγαθών από έδαφος κράτους μέλους επιπροσθέτως θα επιδιώξει να επιτευχθεί συμφωνία με το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ώστε να υιοθετηθεί η απόφαση για τη θέσπιση κοινοτικής δράσης για τις ευρωπαϊκές πολιτιστικές πρωτεύουσες περίοδου 2020-2033 κάτι που έθιξε όπως και το προηγούμενο θέμα η κυρία Πρόεδρος στην εισαγωγή της. Για να επιταχύνει την εφαρμογή της απόφασης για τις ευρωπαϊκές πολιτιστικές πρωτεύουσες η ελληνική προεδρία θα προωθήσει την υιοθέτηση απόφαση για τον ορισμό τη επιτροπή επιλογή και τη εποπτική επιτροπή για το θέμα αυτό. Αυτό ο καθιερωμένος δημοφιλής και με ευρύ αναγνώριση θεσμό. Όπω ξέρετε η πρώτη πολιτιστική πρωτεύουσα ήταν η αθήνα και ήταν μια ιδέα για την οποία δούλεψε πολύ η τότε ε, ελληνίδα υπουργό πολιτισμού μελίνα μερκούρη με τον γάλλο τον τότε γάλλο συναδελφό τη Ζακ Λόγκ αυτός λοιπόν ο δημοφιλής θεσμός αποτελεί βασικό παράδειγμα θετικής συμβολής του πολιτισμού στην μακροπρόθεσμη ευημερία και την αστική και περιφερειακή ανάπτυξη τόσο σε οικονομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Τέλος, η Προεδρία θα προωθήσει την εφαρμογή του πρωτοκόλου πολιτιστικής συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Δημοκρατίας της Κορέας μέσω της υιοθέτησης σχετικών αποφάσεων του Συμβουλίου. Ξέρω ότι έχει γίνει πολλή συζήτηση και ορθώς σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τα θέματα του κινηματογράφου. Θα έχουμε την ευκαιρία στην ανταλλαγή ερωτήσεων και απαντήσεων να συζητήσουμε και αυτά τα θέματα. Απλώς σημειώνω. Σε ό,τι αφορά τον κινηματογράφο έμφαση θα δώσουμε στην ψηφιοποίηση των κινηματογραφικών αιθουσών και της κινηματογραφικής κληρονομιάς και στις νέες πλατφόρμες για τη διανομή όπτικο-ακουστικού και κινηματογραφικού υλικού. Η Ελληνική Προεδρία θα επεξεργαστεί επίσης τη σύσταση του Συμβουλίου για τον Ευρωπαϊκό Κινηματογράφο στην ψηφιακή εποχή υπό την προϋπόθεση ότι θα κατατεθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις αρχές του 2014. Κυρίες και κύριοι, ο πολιτισμός απευθύνεται στην ψυχή και στο νου του ανθρώπου. Ο πολιτισμός επηρεάζει άμεσα τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο γύρω μας. Εάν θέλουμε λοιπόν ο κόσμος μας στο παρόν και στο μέλλον να είναι πιο ανοιχτός, πιο ελεύθερος, πιο δημιουργικός, με λιγότερη δυστυχία, λιγότερες συγκρούσεις και αντιθέσεις, με λιγότερη βία, με περισσότερη δικαιοσύνη, με περισσότερη ανεκτικότητα, τότε ας δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στον πολιτισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι διαπολιτιστικές σχέσεις μεταξύ των λαών μπορεί να γίνουν το προνομιακό πεδίο άβυνσης και επίλυσης των θρησκευτικών και φιλετικών συγκρούσεων διαμορφώνοντας τον καμβά το συνεκτικό ιστό της ειρήνης, της συνεργασίας και της αρμονικής συνύπραξης των λαών. Αυτές είναι οι βασικές σκέψεις που συνιστούν τα κύρια θέματα της ατζέντα της ελληνικής προεδρίας για τον πολιτισμό. Επιτρέψτε μου να παραθέσω κάποιες αντίστοιχες σκέψεις για τον τομέα του αθλητισμού. Ο αθλητισμός Κυρίες και κύριοι, είναι ένας υπέροχος και πολυδιάστατος κόσμος. Κρύβει χαρές, κρύβει ενθουσιασμό, κρύβει νίκες, κρύβει όμως και λύπες, πολλές φορές κρύβει συντριβή και ταπείνωση. Κάποιες στιγμές γίνεται επικίνδυνος και μοιραίος. Τα προβλήματα είναι πολλά, διαπερνούν τα σύνορα και απλώνονται πέρα από αυτά. Κατά συνέπεια, η αντιμετώπιση τους απαιτεί κοινέ πολιτικέ και κοινέ προσπάθειες. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν λείπουν ούτε οι ιδέε, ούτε οι τόλμοι, ούτε οι κοινέ προσπάθειε. Για πρώτη φορά επιχειρήθηκε η προσέγγιση του αθλητισμού στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από προτεραιότητες που εντάσσονται σε συγκεκριμένο πρόγραμμα τριετούς διάρκειας σύμφωνα με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Το πρώτο πρόγραμμα σημείωσε μεγάλη επιτυχία. Η ελληνική προεδρία τώρα έχει την ευθύνη προετοιμασίας και υιοθέτηση του νέου προγράμματος εργασίας για τον αθλητισμό 2014-2017. Είναι ένα έργο υπεύθυνο που απαιτεί συνέχεια και καινοτομία και απαιτεί τη συμβολή όλων σας στη διαμόρφωσή του. Σε κάθε περίπτωση θέλω να υπογραμμίσω ότι σκοπός μου είναι να συνεργαστώ πολύ στενά με τους συναδέλφους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο διάστημα της ελληνικής προεδρίας. Είμαι και εγώ κοινοβουλευτικός τα τελευταία 14 χρόνια και έχω πολύ μεγάλο σεβασμό και πολύ μεγάλη εκτίμηση σε όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από οποιαδήποτε πτέρυγα και αν προέρχονται, οποιαδήποτε και αν είναι η ιδεολογική και πολιτική τους αφετηρία. Το λέω γιατί κανείς δεν βρίσκεται τυχαία εδώ, όλοι είσαστε εντολοδόχοι, όλοι έχετε πάρει εντολή μέσω της ψήφου Ευρωπαίων πολιτών σε ό,τι αφορά τώρα αυτό το δεύτερο πρόγραμμα εργασίας για τον αθλητισμό αποτελεί θα λέγαμε την κατεξοχήν υποχρέωση της ελληνικής προεδρίας η οποία πρέπει να πετύχει μέχρι την 21η Μαΐου του 2014 που έχουμε το Συμβούλιο Υπουργών σχετική συμφωνία. Οι προτεραιότητες που έχουμε θέσει είναι αθλητισμός και κοινωνία, οικονομική διάσταση του αθλητισμού, χρηστή διακυβέρνηση και ακαιρεότητα στον χώρο του αθλητισμού. Εδώ εντάσσονται και η χειραγώγηση των αθλητικών αποτελεσμάτων και ο αγώνας εναντίον του ντόπινγκ. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στον πρώτο άξονα, οι σχέσεις δηλαδή του αθλητισμού με την ευρύτερη κοινωνία, ανήκει το θέμα της ισότητας των φύλων στον αθλητισμό. Μην ξεχνάμε ότι ο αθλητισμός αποτελεί αποτελεσματικότατο μέσο για την ένταξη στην κοινωνία κοινωνικών ομάδων με χαμηλή εκπροσώπηση και συμμετοχή η ελληνική προεδρία θα εστιάσει στο θέμα της βίας που οφείλεται στο φύλλο προστασία των ανηλίκων το οποίο έχουμε επιλέξει ως θέμα του σεμιναρίου που θα γίνει στην Αθήνα στις 20 Μαρτίου. Πρόκειται για ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα που χρήζει νομικού πλαισίου και περαιτέρω παρακολούθησης. Η Ελληνική Προεδρία προτίθεται επίσης να συμμετάσχει στη Διεθνή Διάσκεψη για τη Γυναίκα και τον Αθλητισμό που θα γίνει στη Φιλανδία από τις 12 ως τις 15 Ιουνίου η ελλάδα θέλω να επισημάνω ότι διατηρεί στο κέντρο της προσοχής της το θέμα αυτό και επιδιώκει να συνεισφέρει εμπράκτως στην πρόθεσή του. στη συνέχεια θέλω να τονίσω ότι η ελληνική προεδρία προτίθεται να δώσει ιδιαίτερη σημασία και έμφαση στον αθλητισμό ως πολύτιμο εργαλείο για την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Ο αθλητισμός με τη δυναμική του και τις υποδομές του μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο για την οικονομική ανάπτυξη υπό την προϋπόθεση ότι θα συντονιστούμε καλύτερα θα αξιοποιήσουμε τις υποδομές μας τις εγκαταστάσεις μας θα προγραμματίσουμε εκδηλώσεις κοινού ενδιαφέροντος και θα βγάλουμε μπροστά το έμψυχο δυναμικό μας ως ευρώπη. υπό αυτό το πρίσμα πρέπει να εξετάσουμε τον συντονισμό της χρήσης κληροδοτημάτων των μεγάλων αθλητικών οργανώσεων και αυτό έχει σημασία τώρα που λόγω της οικονομικής κρίσης στην ευρώπη βλέπουμε αρκετές διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις να φεύγουν από την Ευρώπη και να πηγαίνουν προς χώρες οι οποίες αντιπροσωπεύουν τις λεγόμενες αναδυόμενες οικονομίες. Χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Υπήρου. Η Ελλάδα, ε, η ελληνική προεδρία έχει ως σκοπό να διοργανώσει μια ενδιαφέρουσα πολιτική συζήτηση κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου των Υπουργών τον προσεχή Μάιο με θέμα την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα των μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων η ελληνική προεδρία σχεδιάζει το δεύτερο συμπόσιο στην αρχαία ολυμπία κατά το μήνα ιούνιο με το θέμα αυτό. προτείνουμε τη θέσπιση ενός ευρωπαϊκού δικτύου ολυμπιακών εγκαταστάσεων για την εκπεριτροπής διοργάνωση αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων και νομίζουμε ότι δεν υπάρχει καλύτερος χώρος για να συζητήσουμε περισσότερο αυτή την ιδέα από το χώρο του συμποσίου στην αρχαία ολυμπία. ελπίζω κυρία πρόεδρε αξιότιμοι κύριοι και κυρίες ευρωβουλευτές να επιτρέψουν οι υποχρεώσεις σας να είστε κοντά μας σε αυτόν τον θαυμάσιο χώρο τον προσεχή Ιούνιο. Δεν θέλω να κλείσω χωρίς να αναφερθώ σε δύο ακόμη πάρα πολύ κρίσιμα θέματα. Το θέμα της ακαιρεότητος και χρηστής διακυβέρνησης στον αθλητισμό, δηλαδή στην καταπολέμηση των φαινομένων διαφθοράς και στο θέμα της χειραγώγησης των αθλητικών αποτελεσμάτων. Και βεβαίως το θέμα του αντι του αγώνα εναντίον του ντόπινγκ. Θέλω να τονίσω ότι η ελληνική προεδρία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην καταπολέμηση των φαινομένων διαφθοράς στον χώρο του αθλητισμού και ιδιαίτερα στον χώρο των αθλητικών παραγόντων φαινόμενα που έχουν σχέση με το στήσιμο των αγώνων ιδιαίτερα στα θέματα του ποδοσφαίρου. Όπως επίσης δίνουμε ιδιαίτερη σημασία και στην αντιμετώπιση των φαινομένων φάρμακο διέγερσης στον αθλητισμό τα οποία ειλικρινά έρχονται στο φως διαχέονται σε πολύ περισσότερα του ενός αθλήματα και θα έλεγα προκαλούν σοκ στην κοινή γνώμη σε όλους μας από την ευρηματικότητα των μεθόδων που εφευρίσκουν οι πρωταγωνιστές τους προκειμένου να αντιπαρατεθούν στην αξία του εφαγωνίζεστε. Θέλω να σας πω ότι η Ελληνική Προεδρία παρακολουθεί από πολύ κοντά αυτό το αρνητικό φαινόμενο που μας προβληματίζει όλους εν ώψη και της επικείμενης διοργάνωσης των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Σότσι. Σε ό,τι αφορά το ντόπινγκ σας θυμίζω ότι τον περασμένο Νοέμβριο είχαμε στο Johannesburg την τέταρτη παγκόσμια διάσκεψη για τον αθλητισμό κατά την οποία υιοθετήθηκε ο νέος αντιντόπινγκ κώδικας ο οποίος προσφέρει εναρμορισμένες πολιτικές για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο. Κυρίε και κύριοι, η Ελληνική Προεδρία είναι αποφασισμένη να συντονίσει τι προσπάθειες όλων μα προ τη σωστή κατεύθυνση σε στενή συνεργασία με την Γουάντα και με το Συμβούλιο της Ευρώπης. Σας θυμίζω ότι βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την περίοδο η συζήτηση στο Συμβούλιο της Ευρώπης για να έχουμε μια νέα διεθνή σύμβαση, διεθνή συνθήκη για τα θέματα της αντιμετώπισης του ντόπινγκ. Ε, πρέπει να τονίσω ακόμα και κλείνω ότι στις 21 Μαρτίου θα έχουμε στην Αθήνα την άτυπη σύσκεψη διευθυντών αθλητισμού με κεντρικό θέμα την άσκηση και την υγεία αλλά στα πλαίσια των εργασιών της θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και για την σύγχρονη μάστιγα του ντόπινγκ που όπως σας είπα παρουσιάζεται κάτω από διαφορετικές μορφές και με μεγάλη ευρηματικότητα και προβληματίζει ολόκληρο το χώρο του αθλητισμού. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, ευχαριστώ πολύ για την προσοχή και την ανοχή σας. Είμαι στη διάθεσή σας να ακούσω τις σκέψεις σας και να απαντήσω στα ερωτήματά σας. Θέλω με την ευκαιρία αυτή να σας προσκαλέσω την επόμενη Πέμπτη στις 6.30 το απόγευμα στην αίθουσα Μποζάρ των Βρυξελών σε μια εξαιρετική έκθεση που οργανώνουμε εδώ για την εκκίνηση της ελληνικής προεδρίας. Η έκθεση αυτή έχει ως τίτλο «Νοτήλος Navigating Greece» ε, αφορά τη θάλασσα, τη θάλασσα που αποτελεί το συνεκτικό ιστό για όλη σχεδόν την Ευρώπη, τη θάλασσα η οποία μεταφέρει την εμπειρία μας και την παράδοσή μας στις διαφορετικές ιστορικές εποχές και στις διαφορετικές ιστορικές περιόδους. Ε, έχουμε ευρήματα που ορισμένα από τα οποία ταξιδεύουν για πρώτη φορά στο εξωτερικό από σπουδαία ελληνικά μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, αλλά παρουσιάζουμε και την δημιουργία, τις δημιουργίες νέων Ελλήνων οικαστικών καλλιτεχνών για να αναδείξουμε κάτι το οποίο νομίζω είναι δεδομένο για όλη την Ευρώπη, δηλαδή τη συνύπαρξη της ιστορικής παράδοσης με τη σύγχρονη δημιουργία σε όλους τους τομείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Οι συνεργάτες σας είχαν ε, απελπιστεί και ήθελαν να σας πούν για την έκθεση που γίνεται και εδώ ή σήμερα ή αύριο το πρωί. Εγώ πάντως το ανακοίνωσα ότι και εδώ στο κοινοβούλιο μας ε, ε, υπάρχει μια εξαιρετική έκθεση. Ε, αύριο θα γίνουν τα εγγένεια. Αυτό προσπαθούσα να σας πούν, κύριε Υπουργέ, να το αναφέρετε κι εσείς. Το είπα εγώ όπως σας είπα. Ευχαριστούμε. Καλά, εγώ αναφέρθηκα στο Μποζάρ, στην έκθεση του Μποζάρ. Ναι, ναι, ναι, άλλη αυτή του Κοινοβουλίου είναι αύριο. Ναι, και αύριο στο Μποζάρ. Αλλά... Μάρκο Κουρία, πρώτος ομιλητής. Ευχαριστώ και καλώς ήρθε ο υπουργό εδώ. Ευχαριστούμε για όσα μας είπε, τα οποία παρακολούθησα προσεκτικά και με ενδιαφέρον. Αυτό πρέπει να κάνει κανείς όταν ακούμε έναν Έλληνα να μιλά για πολιτισμό. Και κυρίως για όσα είπε για το ότι ο πολιτισμός αποτελεί στρατηγικής φύσεως τομέα και για την Ελλάδα και για την Ευρώπη και σε σχέσεις βέβαια στη σχέση μας με τον υπόλοιπο κόσμο. Σκέφτομαι και ελπίζω ότι αυτό το εξάμεινο θα υπάρξει χώρος και για ένα συλλογισμό, να κάνουμε μία εκτίμηση της πολιτιστικής και καλλιτεχνικής κληρονομιάς και της Ελλάδος και των υπολείπων χωρών της Ευρώπης ολόκληρης που είναι κύριε παράγοντες για να ε, εξάγουμε πολιτισμό πέρα από τα σύνορά μας στον υπόλοιπο κόσμο και η Ελλάδα και η Ιταλία και από εκεί και πέρα θα μπορούσε να υπάρξει μια, ένας σύνδεσμος, μια σχέση πολύ καλή. Και βέβαια θα πρέπει κανείς να ασχοληθεί και με την πρακτική πτυχή. Εσείς αναφερθήκατε σε ένα από τα πρώτα προγράμματα που θα αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Προεδρία για τις Ευρωπαϊκές Πρωτεύουσες Πολιτισμού είναι ένα θέμα που κληρονομάει από άλλα που έχουν γίνει προηγουμένως και από εκθέσεις και εγώ είμαι εισηγητής της έκθεσης για το Κοινοβούλιο και θα πρέπει να σας πω ότι εδώ θα αντιμετωπίσουμε και τις πρώτες δυσκολίες. Σαν Κοινοβούλιο προχωρήσαμε σε μια πρώτη ανάγνωση. Προχωρήσαμε σε μια πρώτη ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο και δεν έκλεισε ακόμα η συμφωνία με το Συμβούλιο όχι για σημαντικά θέματα, όχι για αποκλίνουσες απόψεις επί των πολιτιστικών, όχι για το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο τα έβλεπαν διαφορετικά τα πράγματα, τι σημαίνει σαν αξία αυτή η εμπειρία. Αλλά για κάτι το τυπικό, αυτό μας αναχέτησε. Δηλαδή, ποιος θα πρέπει να ορίζει αυτές τις πολιτιστικές πρωτεύουσες αν το πούμε, το διηγηθούμε εκτός χώρου ε, εδώ μέσα, θα μας πάρουν για τρελούς οι πολίτες μας. Και το Συμβούλιο θέλει να είναι το μοναδικό θεσμικό όργανο που θα πρέπει να καθορίζει τις πόλεις που θα ορίζονται σαν πολιτιστικές πρωτεύουσες Ευρώπης και από την άλλη μεριά όμως η Επιτροπή διαθέτει και Ευρωπαίους εμπειρογνώμονες και εθνικούς που εξετάζουν τις πόλεις αυτές και μετά προτείνουν για να οριστούν αυτές οι πόλεις σαν πρωτεύουσες. Εμείς από την ελληνική προεδρία περιμένουμε ένα άνοιγμα. Αντίθετα όμως, τι παρατηρούμε ότι το πρώτο κείμενο που μας δίνουν είναι ακόμα πιο αυστηρό και άκαμπτο από αυτά που μας αρνήθηκαν ε, το Συμβούλιο άλλους μήνες παλιότερους. Βέβαια θα έχουμε τον τριμερή διάλογο σε λίγο και δεν θα μπω στους δικούς χαρακτήρες αυτών των σημείων, αλλά για ορισμένε πτυχές εμείς επεξεργαστήκαμε λογικές κατά την άποψή μας προτάσεις που λαμβανόταν όλη υπόψη και το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και η Επιτροπή και μας φαινόταν ότι υπήρχε μία σύγκληση για να προχωρήσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα και να βασιστούμε και σε εμπειρογνώμονες και έτσι οι πόλεις και οι πολίτες να μπορούν και εκείνοι να συμβάλλουν για να λάβουμε μία απόφαση σχετικά. Και ολοκληρώνω εδώ για να μπορέσουν να μιλήσουν και οι συνάδελφοι πολύ σωστά είπατε ότι στην ψυχή και στον εγκέφαλο απευθύνεται ο πολιτισμός. Γι' αυτό μην τα δηλητηριάζουμε αυτά. Να δείξουμε ανοιχτό πνεύμα και να λάβουμε μια απόφαση ανοιχτή ακριβώς που να αναγνωρίζει αυτή η απόφαση το δίκαιο όλων να συμμετάσχουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Στην άδελφε Μπόρις. Ευχαριστώ. Και εγώ με αυτή την ευκαιρία θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσίαση που μας κάνατε την παρουσίαση στόχων κοινών. Η Ελλάδα που εκπροσωπείται από εσάς σήμερα είναι μείγμα πολιτισμού και αθλητισμού. Και αν θυμηθούμε την ελληνική φιλοσοφία, ε, νομίζω ότι ε, τους οφείλουμε, οφείλουμε στην Ελλάδα και τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτό είναι μεγάλο επίτευγμα. Στο Βέλγιο είμαστε πολύ πρακτικοί Δηλαδή συνδέουν Υπουργείο Οικονομικών και Αθλητισμού. Άλλο μείγμα πολιτικής αυτό. Όμως πτυχές πολιτισμού και αθλητισμού μπορεί να έχουν τις ίδιες ρίζες, γιατί ο αθλητισμός δεν είναι μόνο ε, ανταγωνισμός και άμυλα, είναι κάτι που βοηθάει να αναπτυχθεί η προσωπικότητα, ιδιαίτερα των νέων και για τις πρωτεύουσες του πολιτισμού, τις πολιτιστικές πρωτεύουσες. Αυτό που είπαμε είναι ότι είναι θετική αυτή η προσέγγιση με τις πολιτιστικές πρωτεύουσες. Θέλουμε λοιπόν οι προοπτικές να διατηρηθούν και στο μέλλον, να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε δηλαδή το θετικό αντίκτυπο των πολιτιστικών πρωτεύουσών και είναι θετικό να μας επιτρέψει ο νέος κανονισμός να τα διασφαλίσουμε αυτά. Είναι πολλές οι πόλεις που επειδή έγιναν πολιτιστικές πρωτεύουσες συνέχισαν να ευημερούν. Η Λίλη στη Γαλλία είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα από πολλά. Γιατί πολλές επιχειρήσεις, πολλές εταιρικές σχέσεις, συμπράξεις αναπτύχθηκαν κατά την περίοδο εκείνη και διατηρήθηκαν μετά. Επίσης, ο ευρωπαϊκός κινηματογράφος, οι ευρωπαϊκές ταινίες, πολύ σημαντικό θέμα. Πριν από δύο χρόνια περίπου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την έκθεσή μου που αφορούσε το μέλλον του κινηματογράφου στην ψηφιακή εποχή. Προφανώς η ψηφιοποίηση είναι πολύ σημαντική, αλλά εξίσου σημαντικό είναι να διασφαλίσουμε ότι θα εφαρμόσουμε πρόγραμμα ε, για τη δημιουργική Ευρώπη με σημαντικούς προϋπολογισμούς και εκεί αναδεικνύεται ο τομέας του κινηματογράφου όχι μόνο σε σχέση με το παρόν αλλά και σε σχέση με μελλοντικές συνεργασίες μεταξύ κρατών μελών. Αν θυμάστε τα πρώτα στάδια αυτού του κινηματογράφου και ε, ο διαγωνισμός θα γίνει φέτος και μπορείτε βεβαίως και εσείς να μας βοηθήσετε να κερδίσουμε και για το νέο διαγωνισμό και βραβείο το, ε, για τη Δημιουργική Ευρώπη ε, υποστήριξη των πολλών. Για τον αθλητισμό θέλουμε και εδώ να έχουμε βέλτιστες πρακτικές το υποπρόγραμμα του Erasmus Συν που αφορά τον αθλητισμό πρέπει να αναπτυχθεί περισσότερο. Ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τους θυμένους αγώνες, ε, που θα, αυτό θα πρέπει να καταπολεμηθεί. Και η Επιτροπή Πολιτισμού και η Νομική Επιτροπή απασχολήθηκαν με το θέμα αυτό. Θα πρέπει να μπορέσουμε να ορίσουμε το αδίκημα καλύτερα, αλλά και τις κυρώσεις που επισύρει ε, ένας θυμένος αγώνας, γιατί προφανώς καταστρέφει όλο το αθλητικό ιδεώδες και ε, κάποιες γενιές που παλιότερα έδειχναν εμπιστοσύνη στον αθλητισμό τώρα βλέπουν να καταραίει το ιδεώδες τους. Θέλω να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία. Ο πολιτισμός είναι πολύ σημαντικό θέμα και νομίζω ότι πρέπει να το συζητάμε ακόμα περισσότερο σε περιόδους κρίσης. Η κυρία Τρούπελ. Ευχαριστώ τον Υπουργό για την παρουσίαση αυτή. Έχω όμως και ένα ερώτημα για τον πολιτισμό και τις εξωτερικές σχέσεις εδώ στην Ευρώπη. Έχουμε αρχίσει να το συζητάμε στο Κοινοβούλιο και ομολογώ ότι δεν έχουμε ακόμη καταλάβει καλά τι ισχύει για την υπηρεσία εξωτερικών σχέσεων της Ένωσης και γι' αυτό θέλω να σας ρωτήσω, γνωρίζετε μήπως εσείς τι συμβαίνει και αν έχετε κανένα πρόγραμμα ή σχέδιο ώστε να σταματήσει επιτέλους αυτή η λεγόμενη πολιτιστική διπλωματία. Μαρή Τερέζ, μαρη τερεζα κύριε Πρόεδρε και τον κύριο Υπουργό για αυτά που μας είπε. Φυσικά οι προτεραιότητες και τα θέματα που μας αναπτύξατε μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα γιατί τα συζητάμε από την αρχή της θητείας μας. Θα σας αναφέρω όμως ένα πιο συγκεκριμένο, τον τομέα της δημιουργίας που έχει μάλλον πολύ μέλλον και είναι ιδιαίτερα σημαντικό να γνωρίζουμε ορισμένους αριθμούς 4,5-5% του ΑΕΠ της Ένωσης πάνω από 8 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης είναι τομέας λοιπόν που ε, αντιπροσωπεύει ακριβώς τη λεγόμενή μας ε, πολιτιστική εξαίρεση. Έλεγα προηγουμένως και στο συνάδελφό σας τον Υπουργό Παιδείας ότι πρέπει να εμφαίνονται όλα αυτά και στον προϋπολογισμό δική σας ευθύνη είναι η επιτήρηση, η εποπτεία των προγραμμάτων που εγκρίνονται ώστε να εφαρμόζονται γρήγορα και αποτελεσματικά αλλά βέβαια και με τον ανάλογη χρηματοδότηση γιατί οι τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας είναι πολύ σημαντικό να χρηματοδοτούνται επαρκώς και να γνωρίζουν όλοι οι δημιουργοί τι ισχύει γιατί πρόκειται για τομέα που δημιουργεί πολλές θέσεις απασχόλησης και αυξάνεται, προοδεύει συνεχώς παρά την κρίση. Ξέρουμε όλοι ότι είναι πολύ ψηλή η ανεργία, διότι πρόκειται για θέσεις απασχόλησης όπου δεν μπορεί να γίνει κατάσταση. Και μάλιστα τα αντίθετα θα έλεγα ότι μπορεί να εξυπηρετήσει ιδιαίτερα περιφέρειες και περιοχές απομακρυσμένες και αυτές. Πρέπει λοιπόν να καταλήξουμε σε χρηματοδότηση και του πολιτισμού και διαρθρωτική, συμπληρωματικά ιδιαίτερα σε περιοχές τουριστικής ανάπτυξης, όπου βέβαια συνδέονται όλα αυτά και με τα θέματα της κληρονομιάς, της πολιτιστικής κληρονομιάς, γιατί και ο πολιτιστικός τουρισμός δημιουργεί ανάπτυξη. Όσο για τον αθλητισμό, Είπατε προηγουμένως ότι η Αθήνα ήταν η πρώτη πολιτιστική πρωτεύουσα. Αυτό γιατί το έθνος σας έχει ιδιαίτερη συμβολική αξία με, την, ε, με τους Ολυμπιακούς κλπ. Αλλά επίσης αξιών τις οποίες συμμεριζόμαστε και εμείς. Και εμείς θέλουμε την ηθική εξυγίανση του αθλητισμού. Ξέρουμε ότι ο αθλητισμός είναι παράγοντας και πολιτιστικής και κοινωνικής συνοχής και αυτό μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Υπάρχουν και άλλα θέματα, τα αναφέρατε, όπως η θέση των γυναικών στον αθλητισμό και ιδιαίτερα το οικονομικό βάρος του αθλητισμού που ξεχνάμε πολλές φορές να το αναφέρουμε και πρέπει να το προωθούμε και αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Παλιαδέλη. Σύντομα όμως παρακαλώ, ε, σύντομα. στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστούμε για την ε, σφαιρική προσέγγιση των θεμάτων που θα σας απασχολήσουν. Ε, να σας θυμίσω ότι ε, κατά πάσα πιθανότητα θα μετέχετε στην απόδοση του πρώτου σήματος Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κληρονομιάς που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε πριν από και θεσπίστηκε νομικά πριν από λίγα χρόνια, στο τέλος του Μαρτίου, αρχές Απριλίου ε, να ευχηθώ ότι θα τον κόπο επί της ελληνικής προεκδρίας να ολοκληρωθεί η διαδικασία που αφορά στην αναδιατύπωση της οδηγίας του 1997 για την παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών και, την επιστροφή του τα κράτη-μέλη και να σας προτείνω ε, δεδομένου ότι στο πρόγραμμα για τη Δημιουργική Ευρώπη που ψηφίστηκε και πάλι ε, που ολοκληρώθηκε μάλλον και ισχύει από το 2007 ως το 2014 η πολιτική κληρονομιά αναφέρεται αλλά στο μέγιστο ποσοστό της και η χρηματοδότηση και ο προγραμματισμός αφορούν περισσότερο το σύγχρονο πολιτισμό. Ελπίζω ότι θα ε, σας προτείνω λοιπόν να αναλάβετε την πρωτοβουλία στο πλαίσιο της, προεδρίας, της να ληφθεί μια απόφαση προκειμένου να προκύψει μια ευρωπαϊκή θέση ό,τι αφορά την μελέτη, την ανάδειξη και τη διαχείριση της πολιτικής κληρονομιάς. Ελπίζω επομένως ως, αντικειμενικό, ως απόλυτο αντικείμενο, όχι στο πλαίσιο του πολιτισμού, αλλά ως ένα αντικείμενο που χρειάζεται ειδική προσέγγιση. Ελπίζω ότι χαίρομαι ότι θα κάνετε δύο συνέδρια με το θέμα αυτό για την πολιτική κληρονομιά και ελπίζω ότι στη διάρκεια τους θα ε, περιμένουμε προσκλήσεις να συμμετάσχουμε και ελπίζω ότι στην ε, διάρκεια τους θα γίνει φανερή και η συμβολή των ερευνητικών κέντρων της Ευρώπης και των πανεπιστημίων της Ευρώπης στην πολιτική κληρονομιά και στην ανάδειξή της. Ευχαριστώ πολύ. I was... I didn't take much of your time, did I? Δεν σας απασχόλησα πολύ καιρό. Λοιπόν, ο κύριος Αγκουράκης και εκείνο σύντομα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, είχα να κάνω μόνο δύο παρατηρήσεις, αν και τα θέματα είναι πάρα πολύ σημαντικά και μεγάλα. Ε, η πρώτη παρατήρηση έχει να κάνει με το ότι κατά την άποψή μου ε, ο πολιτισμός μπορεί να συμβάλλει στον τελικό του σκοπό που είναι πραγματικά η ανύψωση της προσωπικότητας του ανθρώπου και η αναζήτηση καλύτερων κοινωνικών συνθήκων εάν είναι απελευθερωμένος από τα δεσμά και τις, τις, ε, τον εξαναγκασμό της, της εμπορευματοποίησης του χρήματος γιατί είναι προφανές ότι συγκεκριμένα προϊόντα, συγκεκριμένες κατευθύνσεις, συγκεκριμένα έργα προωθούνται ε, εφόσον αυτά επιφέρουν κέρδος. Και από αυτή την άποψη πρέπει να είναι κανείς αρκετά και να έχει και ε, πρόβλημα. Η δεύτερη παρατηρήση που έχω να κάνω είναι ότι η κρίση και όλη αυτή η πολύ δύσκολη κατάσταση, η καπιταλιστική κρίση, έχει οδηγήσει η θελημένα ημί ε, σε αντιπαραθέσεις αν θέλετε. Υπάρχουν δυνάμεις που θέλουν να αντιπαραθέτουν τους λαούς της Ευρώπης μεταξύ τους. Και από αυτή την άποψη ε, έχει μια σημασία κανείς να δει ποια πολιτιστικά προϊόντα και ποιοι πολιτισμοί, ποια πολιτιστικά έργα είναι εκείνα που μπορούν να απαντήσουν σε μια κατάσταση που χειροτερεύει όλο και περισσότερο. Ε, τρίτο ζήτημα έχει να κάνει με την ε, οδηγία για, τα, για τη διαχείριση, για τη συλλογική διαχείριση των δικαιωμάτων ε, πνευματικής ιδιοκτησίας και αυτά τα θέματα δεν έχω υπόψη μου εάν ε, υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, εάν το έχετε στην ατζέντα σας. Πάντως, θα ήθελα να αναφέρω και εδώ ότι υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες ότι όλο και περισσότερο ε, φεύγει από τα χέρια των δημιουργών αυτός ο τομέας, περνά όλο και περισσότερο στον έλεγχο μεγάλων πολυεθνικών ε, εταιριών και το ίντερνετ παίζει εδώ ένα ρόλο. Δημιουργούνται πολύ σοβαρά προβλήματα που εκτός των άλλων περιορίζουν πάρα πολύ την πρόσβαση στον πολιτισμό που και αυτός ο τομέας είναι ένα πολύ σοβαρό ε, επακόλουθο της καπιταλιστικής κρίσης που ζούμε αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ να κάνω μια ερώτηση κύριε Υπουργέ. Ακούσατε ότι η ψηφιοποίηση του κινηματογράφου είναι θέμα πρωταρχικό. Αυτό πώς θα το καταπιαστείτε. Ε, υπάρχει και αναφορά στον προϋπολογισμό νομίζω. Όχι, εμείς προσπαθήσαμε και στην Δημιουργική Ευρώπη να το εντάξουμε. Με τα διαρθρωτικά, μέσω των διαρθρωτικών ταμείων μπορεί να γίνει κάτι. Ε, επίσης, λέτε ότι ο πολιτισμός αφορά και την ψυχή. Συμφωνώ απόλυτα. Αλλά η συμπεριφορά του Συμβουλίου ε, δεν είχε να κάνει με τον πολιτισμό και την ψυχή όταν μίλησε για τις πολιτιστικές πρωτεύουσες για πρώτη φορά. Ε, νομίζω ότι θα πρέπει να ακολουθηθεί μια σωστή διαδικασία εδώ. Υπάρχει μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων και στον τριμερή διάλογο ε, δεχτήκαμε να υπάρξουν δύο ακόμη εμπειρογνώμονες που θα επικουρήσουν το Συμβούλιο και νομίζω ότι εκείνοι πρέπει να μας συμβουλεύσουν. Δεν χρειάζεται δηλαδή η σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου ή του Κοινοβουλίου, γιατί έχουμε τους εμπειρογνώμονες. Δεν είμαστε εμείς, ούτε το Συμβούλιο είναι εμπειρογνώμονες. Θα ήμουν λοιπόν ιδιαίτερα ευγνώμων αν σε εκείνου που στον τριμερή διάλογο ε, ε, αύριο ε, έρθουν να συμμετάσχουν μαζί μας να τους πείτε ότι εδώ παίζει ρόλο και η πολιτισμένη συμπεριφορά από τον πολιτισμό. Ε, μην λέμε όλο εγώ, εγώ. Ούτε εμεί το λέμε αυτό. Αφήστε τους εμπειρογνώμονες να αποφασίσουν και μετά μπορεί να αποφασίσει και ε, η χώρα. Ελπίζω ότι το μήνυμα αυτό θα μπορέσετε να το ε, περάσετε στους ομολόγους σας διότι νομίζω ότι ε, η σκέψη σας είναι σωστή. Ε, αύριο δεν θα είστε βέβαια παρόν, αλλά μπορείτε να επηρεάσετε τους ε, συναδέλφους σας, ούτως ώστε αύριο το αποτέλεσμά μας να είναι καλύτερο. Σας ευχαριστώ πολύ και συγγνώμη για τις πολλές και δύσκολες ερωτήσεις. Α, και η κυρία καμαέβερτε, παρόλο που δεν ήταν γραμμένη στον κατάλογο. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι σύντομη νομίζω. Αν δεν το είχε πει εσύ αυτό που είπες για τις πολιτιστικές πρωτεύουσες θα το έλεγα κι εγώ. Ας τελειώσει πια αυτή η παιδιάστικη συμπεριφορά. Δεν πρόκειται ε, γι' αυτό. Δηλαδή ε, δεν μπορούμε και να τα πούμε έξω τα θέματα που μας απασχολούν και για τα οποία διαπληκτιζόμεθα. Είναι πολύ θετικό ότι το θέμα πολιτισμού και μέσων ενημέρωσης ε, δεν περιλαμβάνεται στο πακέτο με τους Αμερικανούς και το Συμβούλιο μετά από μακρές συζητήσεις μπόρεσε να συμφωνήσει. Και από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών γίνεται προσπάθεια όμως να ξαναμπούν τα θέματα αυτά στις διαπραγματεύσεις. Η ερώτησή μου αφορά αυτό το θέμα. Η ελληνική προεδρία θα είναι στο πλευρό μας, μπορεί δηλαδή να βοηθήσει ούτω ώστε να παραμείνουν τα θέματα μέχρι το τέλος των διαπραγματεύσεων ως έχουν, ώστε ο πολιτισμός να μην περιλαμβάνεται ε, να μην, στις διαπραγματεύσεις. Δεν μιλάμε εδώ για υλικά αγαθά, ε, ε, αλλά άλλα τα οποία δεν θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στις διαπραγματεύσεις. Θα είμαστε πολύ ευγνώμονες αν η ελληνική προεδρία ε, υποστήριζε τη θέση αυτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Minister, please. Κύριε Υπουργέ. Thank Madam καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω και εσάς προσωπικά κυρία Πρόεδρε που λάβατε μέρος στην, ε, στο να θέτετε ερωτήματα, λάβατε μέρος στη συζήτηση με ένα πολύ σημαντικό ερώτημα, αλλά και τους συναδέλφους, κυρίες και κυρίους ευρωβουλευτές, που ε, έλαβαν μέρος στη συζήτηση. Παρακολούθησα όλους με πολύ μεγάλη προσοχή. Γι' αυτό θα επιχειρήσω πολύ γρήγορα, στα πλαίσια του λίγου χρόνου, να κάνω αναφορά σε όλα όσα ετέθηκαν. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ε, κυρίους και κυρίες ευρωβουλευτάς, για τις πολύ τιμητικές αναφορές που έκαναν στην Ελλάδα και στον ελληνικό πολιτισμό διαχρονικά. Ε, εμείς οι Έλληνες, ιδιαίτερα αυτά τα δύσκολα χρόνια της κρίσης, της οικονομικής κρίσης, την οποία θα ξεπεράσουμε με τη βοήθεια και την ελληνική των Ευρωπαίων φίλων και εταίρων μας, αισθανόμαστε περισσότερο Έλληνες, βαθύτερα Έλληνες, αλλά και περισσότερο Ευρωπαίοι και ταυτόχρονα πολίτες του κόσμου. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω όλους τους ε, Ευρωβουλευτάς για τις πολύ τιμητικές αναφορές για την Ελλάδα, για τον ελληνικό πολιτισμό, για τα όσα έχει προσφέρει η Ελλάδα και ο πολιτισμός της στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Ξεκινώ από τον κύριο Σκουρία ο οποίος από ό,τι ξέρω κάνει εξαιρετική δουλειά ως συντονιστής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και ως εισηγητής για τα θέματα των πολιτιστικών πρωτεύουσών. Ε, είναι αλήθεια ότι το θέμα έχει ταλαιπωρήσει αρκετά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ε, θα σας μιλήσω πάρα πολύ ειλικρινά γιατί παρακολούθησα και τον προβληματισμό της Προέδρου της κυρίας Πακ που διαθέτει άλλωστε τεράστια πείρα στα ευρωπαϊκά θέματα και όχι μόνο. Πιστεύω ότι ο τριμερής διάλογος ο οποίος ξεκινάει αύριο αν δεν απατώμε θα αποδώσει και τουλάχιστον ως ελληνική προεδρία είμαστε έτοιμοι να σπρώξουμε τα πράγματα στο να υπάρξει επιτέλους αποτέλεσμα και να κλείσουμε αυτό το θέμα με τρόπο που θα τους ικανοποιεί όλους και αποτελεί ξεχωριστή τιμή για μας γιατί ο θεσμός της πολιτιστικής πρωτεύουσας που πραγματικά απέδωσε και δείχνει πώς μπορεί να διασυνδεθεί ο πολιτισμός με την οικονομία ξεκίνησε η εφαρμογή του από την Αθήνα 1985 Αθήνα πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης έχει στα θεμέλια του τις πρωτοβουλίες όπως σας είπα μιας Ελληνίδας Υπουργού της Μελίνας Μερκούρη αλλά και άλλων εκλεκτών προσωπικότητων από την Ευρώπη όπως θυμήθηκα πριν τον Ζακ Λόγκ. Ε, νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε λύση. Επιμένει η πλειοψηφία του Συμβουλίου ότι θέλει να έχει τον τελευταίο λόγο. Μπορεί να έχει τον τελευταίο λόγο. Δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε από το Συμβούλιο το να έχει τον τελευταίο λόγο. Αλλά οπωσδήποτε τη μεγαλύτερη σημασία την έχει η τελική εισήγηση που θα φτάσει στο Συμβούλιο. Διότι βεβαίως είναι θέμα ε, ενός μιας επιτροπής εμπειρογνωμόνων. Βεβαίως είναι θέμα να υπάρξουν οι ειδικοί οι οποίοι θα μετρήσουν. Μπορεί, μπορεί να προχωρήσει η μία πρόταση, μπορεί να προχωρήσει η άλλη πρόταση. Υπάρχουν υποδομές, υπάρχουν δυνατότητες. Είναι μία σειρά από πάρα πολλά μεγέθη. Είναι πολλές οι παράμετροι που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από περίπτωση σε περίπτωση. Εμείς αισιοδοξούμε ότι θα βρεθεί λύση και είμαστε έτοιμοι να διευκολύνουμε στο να βρεθεί η λύση αυτή. Συμφωνώ ότι στην τελευταία ανάλυση αυτό που έχει σημασία είναι να ακούγονται οι πολίτες. Να ακούγονται οι πόλεις και οι πολίτες. Και να φτάνει η φωνή τους με το σωστό τρόπο στα κέντρα λήψεως αποφάσεων των ευρωπαϊκών θεσμών και της Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τον κύριο Μπόρι. Τον ευχαριστώ επίση για τις τιμητικέ αναφορέ του στην Ελλάδα το θέμα του κινηματογράφου είναι πάρα πολύ μεγάλο, δεν είναι κοντά μας, αλλά καταγράφονται αυτά στα πρακτικά και μπορεί να τα αναζητήσει, γιατί ήταν πολύ σημαντική η τοποθέτησή του. Το θέμα του κινηματογράφου είναι μεγάλο και πρέπει να κάνουμε μια συνολική συζήτηση στην Ευρώπη. Την κάνουμε τη συζήτηση, αλλά πρέπει να διευρυνθεί αυτή η συζήτηση περισσότερο. Ε, έχει σημασία να αναζωογονήσουμε τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο. Έχει σημασία στις ευρωπαϊκές αίθουσες αλλά και στις διεθνείς αίθουσες κινηματογράφου να ακούγονται και να προβάλλονται πάλι ταινίες οι οποίες θα βοηθούν να ακουστούν ευρωπαϊκές γλώσσες. Έχει σημασία να μπορέσει η Ευρώπη να σταθεί με αξιοπρέπεια ανταγωνιστικά στον κινηματογράφο απέναντι για παράδειγμα στις Ηνωμένε Πολιτείες. Ε, η συζήτηση είναι μεγάλη αλλά νομίζω ότι πρέπει να γίνει. Ε, δεν μας ακούει η κυρία Πρόεδρος, γι' αυτό θα κάνω μετά την αναφορά στη συμβολή της στο Erasmus Plus, αλλά θέλω να τονίσω ότι είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι το βραβείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον κινηματογράφο, το, το Lux Prize, το πήρε μια ταινία του Βαν Κρόνιγκεν The broken circle breakdown, νομίζω είναι Βέλγος ο κύριος ε, Βαν Κρόνιγκεν, η οποία διαγωνίζεται για το Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσης ταινίας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι να μην είναι η μοναδική ε, περίπτωση. Ξαναλέω ότι πρέπει να προχωρήσουμε και να διευρύνουμε αυτή τη συζήτηση για τον κινηματογράφο στην Ευρώπη. Πώς η Ευρώπη μπορεί να γίνει και πάλι ανταγωνιστική απέναντι στην αμερικανική κινηματογραφική βιομηχανία, πώς η Ευρώπη μέσα από τον κινηματογράφο μπορεί να προωθήσει γλώσσες, παραδόσεις, δημιουργούς και ούτω καθεξής. Ε, θέλω επίσης να πω, θα κρατήσω την αναφορά μου για το Erasmus Plus όταν γυρίσει η κυρία Πακ, γιατί εκεί θέλω να σημειώσω κάτι πολύ σημαντικό που πέτυχε ίδια. Θα πάω στην κυρία Τρούπελ. Ε, έκανε μια αναφορά στην πολιτιστική διπλωματία και αν δεν κάνω λάθος, αν κάνω θα παρακαλέσω να με διορθώσει, ε, ζήτησε να ξεκαθαριστεί σε επίπεδο Επιτροπής και Συμβουλίου ο ρόλος που μπορεί να έχει η πολιτιστική διπλωματία στις μέρες μας ως εργαλείο της Ευρώπης για τις διεθνείς σχέσεις αλλά και, για τις διαπολιτιστικές σχέσεις. Ε, κοιτάξτε, το είπα στην, ε, στην ομιλία μου ότι θεωρώ πως η πολιτιστική διπλωματία γενικά οι διεθνείς σχέσεις που θα εδράζονται στο πεδίο των διαπολιτιστικών σχέσεων της διαπολιτιστικής επικοινωνίας μπορούν να πετύχουν πολύ περισσότερα από ότι η συνήθις άσκηση διπλωματικής δραστηριότητας σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής. Μπορεί, όπως είπα, να αμβλύνουν φιλετικές συγκρούσεις, θρησκευτικές συγκρούσεις. Η Ελλάδα ανήκει σε μια περιφερειακή ζώνη όπως τα Βαλκάνια, η Μεσόγειος και η Μέση Ανατολή, όπου βλέπουμε να αναζωπυρώνονται και φιλετικές αλλά κυρίως θρησκευτικές συγκρούσεις και να απειλούν την ευρύτερη ειρήνη, σταθερότητα και ασφάλεια στη συγκεκριμένη περιφερειακή ζώνη Λοιπόν, οι διαπολιτιστικές σχέσεις, η πολιτιστική διπλωματία μπορεί να κάνει πολλά και μπορεί να προσφέρει πολλά στην καλή γειτονία, στην ειρηνική συνύπαρξη και στην αρμονική συνεργασία των λαών. Ε, να περάσω στην κυρία Σάντσες ε, Σμιτ. Ε, γνωρίζω ότι είναι η συγγήτρια για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον πολιτισμό. Ε, αποτελεί προτεραιότητά μας να συνδέσουμε περισσότερο τον πολιτισμό ε, με την τρέχουσα οικονομία. Ε, νομίζω ότι τα νούμερα μιλάνε από μόνα τους. Σήμερα περίπου 7 εκατομμύρια πολίτες Ευρωπαίοι ε, έχουν την απασχόλησή τους με τις ευκαιρίες που τους δίνει ο πολιτισμός. αν δεν απατώμε, το ποσοστό συμβολής στο GDP, στο ΑΕΠ είναι περί το 6%. Αυτά μπορούμε να τα διευρύνουμε πολύ περισσότερο. Χρειαζόμαστε συγκεκριμένε πολιτικέ για τι οποίε είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε ω ελληνική προεδρία και για την προώθηση των οποίων είμαστε έτοιμοι να συμβάλλουμε αποφασιστικά. Ε, ο πολιτιστικό τουρισμό βεβαίω αποτελεί ένα πάρα πολύ μεγάλο κεφάλαιο και το ξέρουμε καλά εμεί, οι Έλληνε. Θα σα δώσω απλώ ε, ένα νούμερο ότι σε μια χώρα που έχει 11 εκατομμύρια κατοίκους, πώς είναι η Ελλάδα, για να δείτε τη σημασία που δίνουμε, είχαμε 12 εκατομμύρια επισκέπτες στην πλειονότητά τους ή στην τριπτική τους πλειονότητα ξένοι το καλοκαίρι που μας πέρασε ε, στα ελληνικά μουσεία, στα οργανωμένα ελληνικά μουσεία και στους οργανωμένους ελληνικούς αρχαιολογικούς χώρους. Και μιλάω για οργανωμένους διότι στην Ελλάδα έχουμε 21.000 αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία. Η Ελλάδα είναι ένα απέραντο αρχαιολογικό πάρκο όπως και άλλες χώρες της Ευρώπης και θα υπολογίσετε ότι έχουμε πάνω από 60 εκατομμύρια ογκομετρικά κινητά αρχαιολογικά ευρήματα. Μόνο να σας δώσω ένα, ενδεικτικό νούμερο, μόνο κατά τις εξκαφές για το νέο μετρό της Θεσσαλονίκης, μέχρι σήμερα που συνεχίζονται, έχουμε βρει 150.000 νέα αρχαιολογικά ευρήματα. Κυρίως από τη Βυζαντινή περίοδο, γιατί στη Θεσσαλονίκη έχουμε μια Βυζαντινή πόλη, αστικό οικισμό δηλαδή, κάτω από την σύγχρονη πόλη της Θεσσαλονίκης. Αλλά δεν είναι μόνο η Ελλάδα. Ε, όλη η Ευρώπη είναι διάσπαρτη από αρχαιότητες διαφορετικών ιστορικών περιόδων με τεράστιο ενδιαφέρον. Ναι λοιπόν στον πολιτιστικό τουρισμό, έμφαση στον πολιτιστικό τουρισμό γιατί μπορεί να είναι ένα εργαλείο πολύτιμο για την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Ο αθλητισμός, πολύ σωστά τα είπατε, είναι επίσης σπουδαίος παράγοντας οικονομίας και κοινωνικής συνοχής αλλά πρέπει να αποκαταστήσουμε να συγκροτήσουμε αυτό το δίκτυο συντονισμού και σωστής λειτουργίας των υποδομών που αφήνουν οι μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις. Έχουμε πείρα στην Ελλάδα από αυτό, σε ορισμένε περιπτώσεις και πικράν πείρα της σωστής αξιοποίησης, γιατί μάθαμε, πάθαμε και διορθώνουμε τα λάθη μας για το πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε σωστά σε συνεργασία με τους ευρωπαίους εταίρους και σε συντονισμό με τους ευρωπαίους εταίρους όλες τις υποδομές που διαθέτουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες για θέματα αθλητικών οργανώσεων μετά το τέλος των αθλητικών οργανώσεων με αυτό το δίκτυο σωστής αξιοποίησης και προγραμματισμού εκδηλώσεων. Η κυρία Παλιαδέλη. Πολύ σωστές οι επισημάνσεις. Η κυρία Παλιαδέλη είναι καθηγήτρια αρχαιολογίας όπως ξέρουμε όλοι ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να συμβάλλουμε ως ελληνική προεδρία στην μελέτη ανάδειξη και στη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Και θεωρώ ότι η συμβολή των ερευνητικών και πανεπιστημιακών κέντρων όλων των ευρωπαϊκών χωρών μπορεί και πρέπει να είναι καθοριστική. Σε ό,τι αφορά τον κύριο Αγκουράκη, παρακολουθώ πάντα με πολύ προσοχή τον προβληματισμό του. Ανήκουμε σε δύο διαφορετικές σχολές ιδεολογικές και πολιτικές. Σέβομαι την διαφορετικότητα της άποψής του, αλλά να σας πω κάτι. Δεν θεωρώ το κέρδος κάτι αρνητικό. Χωρίς το κέρδος δεν μπορεί να λειτουργήσει η οικονομία. Άρα το κέρδος είναι θεμητό και επιβεβλημένο. Ο πολιτισμός όμως είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Άλλο αν μπορεί και πρέπει να συνδυάζουμε τον πολιτισμό με την οικονομική ανάπτυξη. Άλλο αν μπορεί και πρέπει ο πολιτισμός να δίνει τη δυνατότητα της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Χωρίς να καθιστούμε τον πολιτισμό πεδίο ασίδωτης κερδοσκοπίας. Γι' αυτό στη σύγχρονη Ευρώπη, στο σύγχρονο κόσμο, στις δυτικές κοινωνίες υπάρχουν κανόνες οι, οποίες, οι οποίοι οριοθετούν τους χώρους της αγοράς και βάζουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο η ιδιωτική οικονομία μπορεί να κάνει τη δουλειά της αλλά η ιδιωτική οικονομία και το κέρδο αποτελούν το μοχλό, την ατμομηχανή για να λειτουργήσουν οι οικονομίες. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ε, τοποθέτηση της κυρίας Πακ, δεν το έκανα ε, πριν γιατί απουσιάσατε, το κάνω τώρα. Θέλω να της αποδώσω τα εύσημα γιατί κατάφερε στο Erasmus Plus να υπάρχει ένας ειδικός προϋπολογισμός για τον αθλητισμό και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και είναι η πρώτη φορά που επιτυγχάνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, αναζητούμε τις δυνατότητες για να μπορέσουμε να έχουμε, αναζητούμε, δεν μπορώ να σας το πω με σιγουριά ακόμη, να μπορέσουν να πληρώσουν τα διαθροτικά ταμεία προγράμματα ψηφιοποίησης κινηματογράφου. Δεν μπορώ να σας απαντήσω με σιγουριά ακόμη. Πρέπει να το αναζητήσουμε. Μακάρι να το καταφέρουμε. Θα είναι κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Σε ό,τι αφορά για τις πολιτιστικές πρωτεύουσες, τοποθετήθηκα κυρία Πρόεδρε ήδη και πιστεύω ότι με την εκκίνηση του τριμερούς διαλόγου, του τριλόγου, θα βρούμε τη σχετική λύση. Ε, τώρα ε, παρακολούθησε επίσης τις ε, τοποθετήσεις της κυρίας Κόμερ που έχει επίσης ρόλο συντονίστριας. δεν διαφωνώ μετά όσα είπατε. Δεν διαφωνώ με τα όσα είπατε ε, συμφωνώ και εγώ ότι πρέπει να τελειώσει αυτή η ιστορία με τα θέματα των πολιτιστικών πρωτευουσών. Ε, το θέμα είναι σύνθετο, δεν είναι απλό. Ε, θα επιμείνω ότι δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε τον τελευταίο λόγο, επαναλαμβάνω, από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αλλά μέχρι να φτάσουμε στο Συμβούλιο που θα έχει τον τελευταίο λόγο, υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία που πρέπει να συμπληρώνεται από ειδικού, από εμπειρογνώμονες, να οριμάζει το θέμα και να καλείται το Συμβούλιο να πάρει την τελική του απόφαση. Εν πάση περιπτώσει δεν θα προκαταλάβω τον τρίλογο, τον τριμερή διάλογο που ξεκινάει αύριο. Η δική μας προσπάθεια θα είναι να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλα τα μέρη να αποφασίσουν και να καταλήξουμε. Θέλω καταλήγοντα να επαναλάβω τον βαθύτατο σεβασμό μου και την εκτίμησή μου προ τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. όπω σα είπα είμαι επί 14 χρόνια Έλληνα κοινοβουλευτικό και την πρόθεσή μου ως ασκούντος την ελληνική προεδρία σε θέματα πολιτισμού και αθλητισμού να συνεργαστώ στενά με όλους σας κυρίες και κύριοι ευρωβουλευτές και βεβαίως με την πρόεδρο της επιτροπής μας για να προωθήσουμε ταχύτατα τα θέματά μας κατά το δυνατόν στο εξάμεινο της ελληνικής προεδρίας. Ευχαριστώ πολύ για την ανοχή και την προσοχή σας. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Μια παρατήρηση αν μου επιτρέπετε δεν πιστεύουμε ότι το Συμβούλιο πρέπει να έχει τον τελευταίο λόγο. Αν κάποιος πρέπει να έχει τον τελευταίο λόγο, είναι Συμβούλιο και Κοινοβούλιο, όχι μόνο Συμβούλιο. Πάνε αυτά. Στη διαδικασία συναπόφασης δεν προβλέπεται πια αυτό. Γι' αυτό δεν νομίζω ότι σε θέματα πολιτιστικών πρωτευουσών πρέπει να επανεισαγάγουμε ένα παλιό θεσμό. Έτσι λοιπόν θα πρέπει νυφάλια να σκεφτούμε αν έχει νόημα να διαπληκτιζόμεθα για το τίποτα. Γιατί ούτε εσείς αποφασίζετε τίποτε, ούτε εμείς. Η Επιτροπή, το ζουρί αποφασίζει. Ε, καλό θα ήταν και θα σας ευγνωμονούσα μέχρι αύριο να βρείτε κύριε Υπουργέ μια λύση όσο γίνεται πιο γρήγορα τέλος πάντων ε, σχετικά με τις ε, επόμενες ε, δύο πολιτιστικέ πρωτεύουσες. Είμαι βεβαία ότι θα μας βοηθήσετε. Ευχαριστώ πολύ και τώρα περιμένουμε τον επόμενο Υπουργό. <laughs> Mr. Kirikoglu. See you. See you in Athens. yes, please instruct your people. Fine. Come, sit you. Ja, es ist kein Mensch mehr da. Niemand mehr da. Was soll ich denn machen? So, can we just continue the... Συνεχίζουμε. Θα ακούσουμε τώρα τον κύριο Κόγλου, υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό, κυβερνητικό εκπρόσωπο, αρμόδιο για τα μέσα ενημέρωσης. Κύριε Κόγλου, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ε, Thank you, Mrs. President. Κυρία Πρόεδρε, είναι ειλικρινά μεγάλη μου χαρά να βρίσκομαι σήμερα εδώ ενώπιον της Επιτροπής σας και να έχω την ευκαιρία να σας παρουσιάσω τις προτεραιότητες της ελληνικής προεδρίας στον τομέα της αρμοδιότητάς μου. Πρωτού προχωρήσω με την παρουσίαση των θεμάτων που θα απασχολήσουν την ελληνική προεδρία στον τομέα των οπτικοακουστικών, θα ήθελα να επισημάνω ότι εν ώψη της διαρκώς αυξανόμενης σύγκλησης των παραδοσιακών με τα νέα οπτικοακουστικά μέσα, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη για περιφρούρηση των βασικών αρχών της ευρωπαϊκής ένωσης που είναι η προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων και ιδίως η ελευθερία της έκφρασης η ανάπτυξη των τεχνολογικών υποδομών και η τήρηση των κανόνων της αγοράς στην ψηφιακή εποχή ο υγιής ανταγωνισμός η διαφάνεια τα ζητήματα αυτά αποτέλεσαν εξάλλου τον κύριο προβληματισμό στις πρόσφατες ευρωπαϊκές διαβουλεύσεις τα αποτελέσματα των οποίων θα μας δείξουν τις κατευθύνσεις στις οποίες θα πρέπει να κινηθούμε. Γνωρίζουμε τη μακροχρόνια προσπάθεια του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περαιτέρω προώθηση της ελευθερίας, της έκφρασης και της πολυφωνίας των μέσων στην Ευρώπη περαιτέρω είναι γνωστό ότι με την ψηφιακή ατζέντα και τη στρατηγική της ευρωπαϊκής ένωσης για την επίτευξη της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης μέσω των νέων ψηφιακών τεχνολογιών επιχειρείται η ρυθμιστική ενοποίηση των εθνικών οπτικοακουστικών αγορών των κρατών μελών. στα περισσότερα κράτη μέλη συμπεριλαμβανομένης και της χώρας μου οι νέες υπηρεσίες καταλαμβάνουν ήδη ένα σημαντικό μέρος της εθνικής οπτικοακουστικής αγοράς στο πλαίσιο αυτό εκτιμούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να διασφαλιστεί η δυνατότητα πρόσβασης σε όλες τις νέες πλατφόρμες και υπηρεσίες από όλους και να εξασφαλιστεί η ελεύθερη ροή πληροφοριών στην εσωτερική αγορά με την άρση των εμποδίων εισόδου νέων παικτών στην αγορά και την ενίσχυση της διαφάνειας. Και τώρα θα σας παρουσιάσω τα θέματα που θα απασχολήσουν την ελληνική προεδρία στον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων, τα οποία είναι τα εξής. Πρώτον, υιοθέτηση νέας απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την υπογραφή εκ μέρους της Ένωσης της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την νομική προστασία των υπηρεσιών που βασίζονται ή συνίστανται σε πρόσβαση υπό όρους του Συμβουλίου της Ευρώπης σε συνέχεια της έκδοσης της ε, από 22 Οκτωβρίου του 2013 σχετικής απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ανωτέρω απόφαση του δικαστηρίου της ευρωπαϊκής ένωσης κρίθηκε ότι η υπογραφή και η επικύρωση της ευρωπαϊκής σύμβασης του συμβουλίου της ευρώπης για την νομική προστασία των υπηρεσιών που βασίζονται ή συνίστανται σε πρόσβαση υπό όρους δεν αποτελεί συντρέχουσα αρμοδιότητα της ευρωπαϊκής ένωσης και, και των κρατών μελών αλλά αποκλειστική αρμοδιότητα της ευρωπαϊκής ένωσης προκειμένου να εφαρμοστεί η απόφαση του δικαστηρίου της ευρωπαϊκής ένωσης θα πρέπει να εκδοθούν δύο νέες αποφάσεις του συμβουλίου για την υπογραφή και την επικύρωση της ευρωπαϊκής σύμβασης του συμβουλίου της ευρώπης. στο πλαίσιο αυτό η ελληνική προεδρία θα επιδιώξει την έγκριση νέας απόφασης του συμβουλίου για την εκ μέρους της ένωσης υπογραφή από την ευρωπαϊκή επιτροπή της εν λόγω σύμβασης του συμβουλίου της ευρώπης έως τα μέσα απριλίου του 2014 προκειμένου να τηρηθεί η εξάμεινη προθεσμία που έχει θέσει το δικαστήριο της ευρωπαϊκής ένωσης. οι σχετικές εργασίες του συμβουλίου θα βασιστούν εκ νέου στις αντίστοιχες αρχικές προτάσεις της ευρωπαϊκής επιτροπής που είχαν υποβληθεί το 2010 και τις οποίες η ελληνική προεδρία έθεσε ήδη στα κράτη μέλη κατά την πρώτη συνεδρίαση της ομάδας οπτικοακουστικών θεμάτων του συμβουλίου στις 17 Ιανουαρίου επισημαίνεται ότι η δεύτερη απόφαση του συμβουλίου για την επικύρωση της εν λόγω σύμβασης θα πρέπει να εκδοθεί μελλοντικά με τη συμμετοχή του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου βάσει της διαδικασίας επικύρωσης διεθνών συμβάσεων. δεύτερο θέμα είναι η επεξεργασία των αποτελεσμάτων των τριών ευρωπαϊκών διαβουλεύσεων σχετικά με η πρώτη αφορά την προώθηση της ανεξαρτησίας των ρυθμιστικών αρχών που είναι αρμόδιες για τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες η δεύτερη διαβούλευση αφορά την προετοιμασία για την πλήρη σύγκληση στον οπτικοακουστικό κόσμο, Connected TV, οικονομική μεγέθυνση, δημιουργία και αξίες και τρίτο την προώθηση της ελευθερίας της έκφρασης και της πολυφωνίας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνέχεια της πρώτης έκθεσης για την εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, διεξήγαγε το περασμένο έτος δύο ευρωπαϊκές δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με την προώθηση της ανεξαρτησίας των εθνιστικών αρχών που είναι αρμόδιες για τα οπτικοακουστικά και για την προετοιμασία για την πλήρη σύγκληση στον οπτικοακουστικό κόσμο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ολοκλήρωσε επίσης κατά το έτος 2013 την Ευρωπαϊκή Δημόσια Διαβούλευση σχετικά με την προώθηση της ελευθερίας της έκφρασης και της πολυφωνίας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης η ελλάδα συμμετείχε ενεργά σε όλες αυτές τις ευρωπαϊκές δημόσιες διαβουλεύσεις κινητοποιώντας με κάθε τρόπο τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς προκειμένου να διατυπώσουν τις απόψεις τους και στη συνέχεια συνεισέφερε με εμπεριστατωμένες απαντήσεις και στις τρεις διαβουλεύσεις λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις των διαφερομένων εθνικών φορέων. Στόχος της ελληνικής προεδρίας είναι του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να εργαστεί επί των αποτελεσμάτων των ανωτέρων διαβουλεύσεων, η δημοσίευση των οποίων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να αναπτύξει μεταξύ άλλων και έναν επικοδομητικό διάλογο μεταξύ των κρατών μελών για το λόγο αυτό η ελληνική προεδρία του συμβουλίου της ευρωπαϊκής ένωσης θα ενθαρρύνει την ενημέρωση σχετικά με τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων η οποία μπορεί να γίνει τμηματικά και σταδιακά εκ μέρους της ευρωπαϊκής επιτροπής σε συνάρτηση με την πορεία της ανάλυσης των απαντήσεων που έχει λάβει από τα κράτη μέλη της ευρωπαϊκής ένωσης. Ευελπιστούμε δε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορέσει να παρουσιάσει συνολική ανάλυση των αποτελεσμάτων των διαβουλεύσεων στο Συμβούλιο Υπουργών του Μαΐου 2014. Τέλος, θα ήθελα επίσης να σας ενημερώσω για μια σημαντική διοργάνωση στον τομέα των οπτικοακουστικών, η οποία θα πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο στην Αθήνα στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου. Αντιλαμβανόμενοι τις σημαντικές προκλήσεις που ανακύπτουν από τη σύγκληση των παραδοσιακών μέσων με τα νέα οπτικοακουστικά μέσα και ιδίως τον παγκόσμιο και πολυσύνθετο χαρακτήρα του διαδικτύου αλλά και τη δημιουργία νέων υπηρεσιών και συσκευών θα επιδιώξουμε στο πλαίσιο της ελληνικής προεδρίας τη συνέχιση του πολιτικού διαλόγου που ξεκίνησε η λιθουανική προεδρία. Ειδικότερα θα επιδιώξουμε τη διεξοδική εξέταση των ζητημάτων που ανακύπτουν από την ηλικιώδη μεταβολή του οπτικοακουστικού πεδίου με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των ανηλίκων στην ψηφιακή εποχή. Στο πλαίσιο αυτό, η Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης της ελληνικής κυβέρνησης θα διοργανώσει στις 14 και 15 Απριλίου του 2014 στην Αθήνα διάσκεψη με θέμα «Η προστασία των ανηλίκων στην ψηφιακή εποχή», στην οποία θα κληθούν να συμμετάσχουν εκπρόσωποι των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συμβουλίου της Ευρώπης και άλλων διεθνών οργανισμών των δημοσίων διοικήσεων των ευρωπαϊκών κρατών των ρυθμιστικών αρχών της ακαδημαϊκής κοινότητας και των ενδιαφερομένων φορέων της αγοράς. Στην ελόγω διάσκεψη προγραμματίζεται η ένταξη, μεταξύ άλλων, των παρακάτω θεματικών ενωτήτων. Προστασία των ανηλίκων σε σχέση με την Connected TV, το διαδίκτυο, τη διαφήμιση, τις εμπορικές ανακοινώσεις λιπαρών τροφών, την ελευθερία της έκφρασης, την παιδεία στα μέσα ενημέρωσης. Ευελπιστούμε για τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διάσκεψη. Γνωρίζουμε ότι τις μέρες εκείνες συνεδριάζει η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα είναι και η τελευταία συνεδρίαση της τετραετίου της θητείας του. Ωστόσο σας προσκαλούμε, εάν μπορείτε, να συμμετάσχετε στη διάσκεψη για την παρουσία της Επιτροπής σας και καθενός από εσάς θα προσδώσει ιδιαίτερο κύρος και ενδιαφέρον στη διάσκεψη. Και φυσικά κάθε πρόταση είναι ευπρόσδεκτη σε σχέση με τον εμπλουτισμό της θεματολογίας. Θα ήθελα επίσης να σας διαβεβαιώσω ότι η χώρα μου ως Προεδρεύουσα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιθυμεί να συνεχίσει την καλή συνεργασία του Συμβουλίου με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο πεδίο των οπτικοακουστικών θεμάτων, γνωρίζοντας ότι η προώθηση των δημοκρατικών αρχών και των πολιτιστικών αξιών αποτελεί κοινό μας στόχο. Και θα ήθελα τέλος να σας διαβεβαιώσω ότι θα θέλαμε να είναι ανοιχτός ο διεύλος επικοινωνίας με την Επιτροπή σας. Σας ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε θερμά. Ο κύριος Παπα-Νικολάου ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, καλώς ήρθατε. Δυστυχώς είστε ο τελευταίο σήμερα που κάνετε την εισήγηση και γι' αυτό βλέπετε ότι πολλοί συνάδελφοι απουσιάζουν. Είχαμε και παράλληλες άλλες ακροάσεις, άλλες επιτροπές και ε, αυτό δεν είναι πάντα εύκολο για μας, ξέρετε, να πηγαίνουμε και να ερχόμαστε. Ε, και από την πολιτική μας ομάδα δεν είναι σήμερα μαζί μας οι συνάδελφοι που ασχολούνται πιο πολύ με τα ακουστικά μέσα, έχουν δώσει περισσότερη έμφαση στα θέματα αυτά και έχουν κάνει σχετικές εκθέσεις. Ε, είναι εδώ βέβαια η κυρία Κάμεβερτ και, και η κυρία Κώστα έχει ασχοληθεί. Ε, φαντάζομαι θα ρωτήσουν και εκείνες. Ε, η δική μου ερώτηση είναι η εξής. Ε, κουβεντιάζουμε για τα οπτικοακουστικά μέσα και κουβεντιάσαμε προηγουμένω προηγούμενε ενότητε και με τον Υπουργό Παιδεία και ε, τον κύριο Παναγιοτόπουλο σε σχέση με τι ευκαιρίε που δίδονται ε, από του πυλώνε αυτή τη ε, Επιτροπή για ανάπτυξη, για δημιουργία νέων θέσεων εργασία, για ευκαιρίε ιδιαίτερα στου νέου ανθρώπου. Τα οπτικοακουστικά μέσα λοιπόν δίνουν τέτοιε ευκαιρίε τα οπτικοακουστικά μέσα δεν είναι μόνο τα παραδοσιακά που ξέραμε μέχρι σήμερα. Συζητάμε πλέον και για τα ψηφιακά οπτικοακουστικά μέσα και τι νέε κατευθύνσει, τι νέε πλατφόρμε, τι δυνατότητε που δίνουν νέε τεχνολογίε. Αναφερόμαστε συνεχώ εδώ στην Επιτροπή μα στην ψηφιακή εποχή. Ε, λοιπόν πώ η ελληνική Προεδρία θα μπορέσει στο σύντομο χρόνο που έχει να δώσει έμφαση στα ζητήματα αυτά, πώ ο τομέας των οπτικοακουστικών μέσων όπως σήμερα διαμορφώνεται και όπως σήμερα αναπτύσσεται μπορεί να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες ιδιαίτερα για τους νέους της Ευρώπης. Σας ευχαριστώ πολύ. Uh, κυρια Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ θερμά κύριε Υπουργέ για αυτά που μας είπατε. Δύο παρακλήσεις θέλω να εκφράσω. Δεν είναι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ακόμα και κατά το παρελθόν δεν ασχολήθηκε εντατικά με θέματα οπτικοακουστικής ε, πολιτικής ε, και μέσων και τώρα πάλι το κάνει και υπενθυμίζω την ευρεία πλειοψηφία ε, υπέρ του Connected TV, την έκθεση πρωτοβουλίας όπου είχαμε προσθέσει πολλά πράγματα και είχαμε πει ότι θα πρέπει να υπάρξει κάποια αναθεώρηση της οδηγίας για τα οπτικοακουστικά και η Κομισιόν θα πρέπει να το σκεφτεί αυτό. Νομίζω ότι δεν πρέπει να επανεφευρίσκουμε τον τροχό κάθε φορά όσοι ασχολούνται με το θέμα, αλλά να ανατρέχουν στις ιδέες που είχε κατά καιρούς αναπτύξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τέλος, μια άλλη παράκληση ε, σε σχέση ε, με τις ψηφοφορίε που είχαμε σήμερα το πρωί. Μεγάλη πλειοψηφία σε αυτή την Επιτροπή σήμερα το πρωί ψηφίσαμε το σχέδιο έκθεσης για την ψηφιακή εσωτερική αγορά με πολλές τροποποιήσεις σε σχέση με το, πρόγραμμα, το σχέδιο της Κομισιόν και θέλουμε να υπάρχει νομική διασφάλιση της ουδετερότητας των ε, δικτύων, να υπάρχει η αρχή του best effort ε, νομοθετημένη, ε, η εξειδικευμένες υπηρεσίες specialized services ε, να υπόκεινται ε, σε συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ούτω ώστε να έχουμε κατάλληλες πρακτικές ε, και στην διαδικτυακή εποχή. Θα πρέπει δηλαδή να ξέρουμε πού θα υπάρχει και που δεν υπάρχει πρόσβαση. Θέλουμε σε αυτό την υποστήριξή σας. Θα χρειαστούμε όλη την υποστήριξη που μπορούμε να έχουμε, γιατί αυτό το θέμα δεν ε, εκτοξετάζουν μέσα από την πολιτιστική πολιτική, αλλά και μέσα από τη βιομηχανική πολιτική. Και πολλές φορές εκεί τα επιχειρήματα διαφοροποιούνται. Εσείς ως υπουργό υπεύθυνο για τα ε, μέσα ενημέρωσης στο Συμβούλιο ε, θα θέλαμε να υποστηρίξετε το θέμα αυτό, να μην εξετάσουν το θέμα μόνο μέσα από τη σκοπιά της βιομηχανίας, αλλά και των επιπτώσεων που θα υπάρχουν από τα ε, μέσα ενημέρωσης, ε, ούτως ώστε να υποστηριχθεί το, η Επιτροπή Πολιτισμού και να ε, προσελκύσουμε και επίσης και την κοινή γνώμη στο σημαντικό αυτό θέμα. Ευχαριστώ. Κύριε Κώστα. Κύριε Υπουργέ, σας εύχομαι και εγώ καλή δουλειά και ευχόμαστε η Ελληνική Προεδρία να δημιουργήσει να ανοίξει καινούριο δρόμο και στα θέματα του πολιτισμού, επικοινωνίας κλπ. μέσω των καταλληλοπρογραμμάτων προγραμμάτων όπως ήδη ακούσαμε στην παρουσίαση. Πολύ με ενδιαφέρουν αυτό που είπατε εσείς ότι θα πρέπει κανείς να καταλάβει ότι για την παρασκευαστική εργασία για να ασχοληθούμε με τα οπτικοακουστικά μέσα και την οδηγία γιατί τις διαβουλεύσεις ε, μέσω της Επιτροπής και τώρα τα πρόσφατα ψηφίσματα του, όπως είπε η Ρέβερτ, του Κοινοβουλίου έφτασε η στιγμή να κάνουμε ένα βήμα προς τα εμπρός προς την κατεύθυνση αυτή. Θα ήθελα να σας πω ότι σχετικά με τις διαβουλεύσεις που υπενθυμίσατε για τα οπτικοακουστικά μέσα, για τηλεόραση, για την ελευθερία έκφρασης και την, το θέμα των αρχών. Μετά από τα αποτέσμα της διαβούλευσης θα πρέπει να ξεκινήσουμε την όλη διαδικασία και να επιταχυνθεί η εφαρμογή αυτών των στόχων, η υλοποίησή τους. Εμείς ε, ε, ακριβώς υπογράψαμε μια αναφορά των Ευρωπαίων πολιτών πάνω σε αυτά για να μπορέσει κανείς να κάνει κάτι το περισσότερο, το ισχυρότερο σχετικά με τον πλουραλισμό των ε, ε οπτικοκουστικών μέσων και ε, τη μη συγκέντρωση εξουσίας και διοκτησίας τηλεόρασης ε, κλπ. Χρειάζεται προσοχή αυτά και χαίρομαι για την πρωτοβουλία σας για να συμμετάσχουν ε, για την συμμετοχή των ανηλίκων σε αυτή την ψηφιακή εποχή. Και εδώ το Κοινοβούλιο το είχε πει αυτό, ότι ήθελε να προχωρήσει κάπως περισσότερο στη σημερινή κατάσταση. Και είδαμε και τη σύσταση της Επιτροπής σε αυτό το πεδίο, σε αυτό το τομέα. Αλλά ορισμένα αιτήματα σε αυτήν το θέμα να μπορέσουν να ενταχθούν και σε εθνικές νομοθεσίε Κάτι σχετικά με τις ταινίε σχηματογραφικές. Το είπε και ο συνάδελφός σας πριν. Και η κυρία Πάκ επίσης το είπε με τον συνάδελφό σας, τον Υπουργό Πολιτισμού. Χαίρομαι που μιλάτε για αυτά, γιατί εδώ στην Επιτροπή αντιμετωπίζουμε πολλές δυσκολίε για να καταλάβουν ότι αυτό το αρχείο το κινηματογραφικό όπως επίσης και της κληρονομιάς γενικά της κινηματογραφικής. Δεν είναι ένα θέμα που αφορά μόνο εθνικό επίπεδο και τα διαφορετικά ταμεία ε, στην Ευρώπη ε, ο προϋπολογισμός δεν είναι ο κατάλληλος, δεν είναι επαρκής. Θα πρέπει να εργαστούμε περισσότερο από τη στιγμή που έχετε παρόμοια πρόθεση, γιατί νομίζουμε ότι δίνουμε μάχη στο Κοινοβούλιο. Να υπάρξει αυτή η δυνατότητα ψηφιοποίησης και όλα αυτά να εφαρμοστούν στην ονειρομιά έτσι την κλιματογραφική θα πρέπει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο να υποστηριχθεί και όχι μόνο σε εθνικό. Στα σχέδια αυτά ορισμένα προχωρούν, θα πρέπει να διευρυνθούν κανονικά για την ψηφιοποίηση και των αρχείων των κλιματογραφικών ε, σε αυτό. Δεν έχουμε πάντα μια ενιαία βέβαια απάντηση από ορισμένου επιτρόπου που λένε ότι η κληρονομιά αυτή η κλιματογραφική αφορά μεμονωμένα κράτη. Αυτά και ευχαριστώ. Είναι ενδιαφέρον κατά την απόψη μου. Κυρία Τρούπελ, ευχαριστώ. Ευχαριστώ και για αυτά που είπατε και για όλη σας την παρουσίαση. Θα ήθελα να συμπληρώσω μερικά πράγματα σε αυτά που ακούστηκαν. Το θέμα δηλαδή των δημοσίων σταθμών τηλεοπτικών, δημοσίων ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών. Αυτά είναι δημόσια αγαθά και Υπάρχει η σύμβαση της UNESCO για την πολιτιστική ποικιλομορφία. Είναι φανερό ότι οι δημόσιοι σταθμοί έχουν εκτός από επιχειρήσεις είναι και μεταφορείς περιεχομένων και μηνυμάτων. Επομένως, η λεγόμενη ουδετερότητα του ίντερνετ Υπάρχει και γι' αυτό πρέπει και εμείς να υπενθυμίσουμε ότι και η ελληνική προεδρία πρέπει να παίξει έναν σαφή ρόλο και έχει αυτό, σε αυτό το θέμα. So, last but not least, Mr. Angouraki. Τέλος ο κύριος Αγκουράκης. Πρόεδρε, ε, είναι μια σημαντική συζήτηση. Δυστυχώς εγώ δεν έχω την τιμή να συμμετέχω, όπως ξέρετε, σε αυτή την Επιτροπή. Εκ μέρους της ομάδας αριστεράς δεν είναι εδώ η συγκήτριά μας. Εν πάση περιπτώσει, ορισμένες σκέψεις ε, με βάση τα όσα ακούσαμε τον κύριο Υπουργό. Καταρχήν, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινεί, το λέω με όλη την ε, υπευθυνότητα που μπορώ να έχω, δεν υπάρχει ελευθερία έκφρασης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτή είναι η αλήθεια. Κυρία Πρόεδρε, είχαμε μία αντιπαράθεση πριν σε σχέση με το κοινωνικό σύστημα, με τους επιχειρηματίες και τον καπιταλισμό. Και όταν λέω ότι δεν υπάρχει ελευθερία έκφρασης, λέω το εξής. Βεβαίως υπάρχουν οι επιχειρηματίες διότι είναι καπιταλιστικό το σύστημα. Αλλά όπως αγνωρίζετε άριστα, και αυτό αφορά και την εκπαίδευση, οι επιχειρηματίες είναι η ελάχιστη μειονότητα σε αυτό το σύστημα που υπάρχει. Και τις αξίες και την παραγωγή την παράγουν οι εργάτες, οι εργαζόμενοι. Ε, λοιπόν, οι εργαζόμενοι δεν έχουν άποψη. Δεν έχουν θέση στην ε, τηλεόραση. Είτε δημόσια είναι αυτή, είτε ιδιωτική. Δεύτερο, ε, και βέβαια και πολιτικά κόμματα πάρα πολλά πολιτικά κόμματα. Η κατάσταση στην Ελλάδα είναι δραματική. Δεύτερο ζήτημα, στην Ελλάδα μεγάλος, ε, μεγάλο μέρος της, του τηλεπτικού προϊόντος, των τηλεπτικών εκπομπών είναι ιδιωτικές. Η ποιότητα σας πληροφορώ. Το περιεχόμενο των εκπομπών είναι απαράδεκτη. Απαράδεκτη από κάθε άποψη. Και πολιτιστική και μορφωτική και αισθητική, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Αλλά το ίδιο ισχύει και για τη δημόσια τηλεόραση. Σε λιγότερο βαθμό βέβαια, αλλά ισχύει. Και για το περιεχόμενο δεν γίνεται καμία συζήτηση. Αυτό που συζητάμε είναι ρυθμίσεις, είναι απελευθέρωση, είναι αγορά, είναι ψηφιακά, είναι... με το περιεχόμενο τι θα γίνει. Θα συνεχίσει να είναι αυτό το άθλιο περιεχόμενο το οποίο βεβαίω είναι συγκεκριμένο γιατί γίνεται. Διότι χρειάζεται να υπάρχει μια συγκεκριμένη πλήση εγκεφάλου. Όπως πλήση εγκεφάλου γίνεται τα τελευταία 4-5 χρόνια και με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τις πολιτικές που εφαρμόζονται σε βάρος των εργαζομένων σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είτε δημόσια είναι αυτά, είτε, είτε ιδιωτικά. Ε, δεν υπάρχει αντίθετη άποψη, δεν υπάρχει αντίθετη γνώμη, δεν υπάρχει άποψη που λέει ότι πρέπει ο κόσμος να αντισταθεί, να οργανωθεί, να παλέψει. Αυτό δεν υπάρχει, είναι, είναι απαγορευμένη άποψη. Και τελευταία βέβαια δεν είναι τυχαίο ότι συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Όπως γνωρίζετε και θα έπρεπε κατά τη γνώμη μου η Επιτροπή σας και γενικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αντιδράσει πολύ πιο δυναμικά και πολύ πιο συγκεκριμένα. Στην ουσία συγκάλεψε αυτό το απαράδεκτο που έγινε το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Η κυβέρνηση με μια ε, αυταρχική απόφαση να κλείσει τη δημόσια τηλεόραση να εξαφανιστούν από, τα, από τις οθόνες οτιδήποτε, να είμαστε μήνες με μια μαύρη οθόνη και βεβαίως η πλειοψηφία του Ευρωκοινοβουλίου, τελειώνω κυρία Πρόεδρε, γιατί, γιατί ενοχλείστε, αυτές είναι αλήθειες κυρία μου. Και αυτές οι αλήθειες πρέπει να υποθούν, θα πάμε σε ευρωεκλογές, θα κριθούμε όλοι για το τι κάναμε και το τι είπαμε. Και εμείς που μιλάμε και αυτοί που δεν μιλάνε. Λοιπόν, αυτό αποτέλεσμα ήταν να αναπολυθούν 2.500 εργαζόμενοι, να, να χειροτερέψει ακόμα περισσότερη η κατάσταση και να γίνεται ακόμα πιο άθλια η δημόσια τηλεόραση στην Ελλάδα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, Αγαπητέ συνάδελφε Αγγουράκη, αναφερθήκατε σε μένα. Εγώ, ναι, είπα κάτι, ανέφερα κάτι ως πρόεδρος Ντόρις ε, Πακ. Θέλω να πω ότι Τρεις φορές είχατε τη δυνατότητα επιμακρών να μας κοινοποιήσετε την άποψή σας ε, αυτά. Όχι, δεν ήταν δική σας, ε, δεν δώσατε εσείς αυτή τη μάχη. Ε, απαντάει σε παρέμβαση εκτός μικροφώνου. Λοιπόν, πολλές φορές μας τα είπατε, ωραία και καλά. Μπορείτε να τα βάλετε και στο, στην ιστοσελίδα σας για να τα ξέρουμε. Εν μέρη έχετε δίκιο, σε μεγάλο βαθμό έχετε άδικο, όμως εγώ τώρα δεν τολμώ να μπω στη, στα ελληνικά δεδομένα. Θέλω να δώσω τον ε, λόγο στον Υπουργό, ο οποίος θα απαντήσει στις ερωτήσεις που του έγιναν. Παρακαλώ κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, να τα πάρω με τη σειρά. Πρώτα τον κύριο Παπα-Νικολάου. Ε, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, προτεραιότητες, προτεραιότητες που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το εξάμεινο που η Ελλάδα έχει την Προεδρία του Συμβουλίου είναι η, απασχόληση, η ανάπτυξη και η απασχόληση. Είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας. Αυτή τη στιγμή ο χώρος, οι τεχνολογικές εξελίξεις στον χώρο των οπτικοακουστικών μέσων προσφέρει τις δυνατότητες για να παλέψουμε και εκεί το τέρας της ανεργίας. Είναι ο μεγαλύτερος εχθρός μας, είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά είναι και ο, ο μεγαλύτερος εχθρός μας στην Ελλάδα. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι στην Ελλάδα χτυπηθήκαμε από την ανεργία όπως καμία άλλη χώρα. Έχουμε τεράστια ποσοστά, ιδιαίτερα στους νέους, είναι αγγίζει το 60% είναι ένα εφιαλτικό νούμερο και ταυτόχρονα έχουμε νέους με δεξιότητες. Νέους με δεξιότητες, νέους καταρτισμένους και νέους που ιδιαίτερα στον χώρο των οπτικοακουστικών μέσων έχουν πολλά να προσφέρουν. Λοιπόν, αυτές οι κατευθύνσεις που έχει δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και που σκοπεύουμε να προωθήσουμε σαν Ελληνική Προεδρία δημιουργούν τη δυνατότητα αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών. Η, όπως ανέφερα στην εισήγησή μου, η δυνατότητα ευκολότερης πρόσβασης σε όλους τους παίκτες, η δυνατότητα για παράδειγμα μια ομάδα νέων δημιουργών να μέσω μιας πλατφόρμας των νέων υπηρεσιών να μπορέσει να έχει άμεση πρόσβαση στο κοινό και να μην χρειάζεται την έγκριση κανενός καναλάρχη κυρία Γκουράκη, να μην υπάρχουν ε, οι λιγότεροι δυνατοί περιορισμοί, αλλά θα απαντήσω εκτενέστερα σε αυτά που είπατε αργότερα. Ε, εκεί λοιπόν, στον χώρο των οπτικοακουστικών μέσων, συνδυασμένοι οι Ευρωπαίοι μπορούν να φέρουν αποτελέσματα. Κάθε μία χώρα είμαστε μία μικρή αγορά, αλλά όλοι μαζί είμαστε μία μεγάλη. Η διασύνδεσή μας είναι επιτακτική σημασίας. Ε, και ελπίζουμε, πιστεύω ειλικρινά, γιατί είμαι και εγώ από το χώρο, είμαι δημοσιογράφος κατ' επάγγελμα, είμαι, ε, και δούλεψα κοντά 20 χρόνια στον χώρο των μέσων ενημέρωσης. Ε, γνωρίζω πολύ καλά ότι, για παράδειγμα, και επίσης οι δημοσιογράφοι, να ξέρετε, στην Ελλάδα έχουν από τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας. Αγγίζουν, ε, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΥΕΑ, σχεδόν τα μισά μέλη του, της Ένωσης Συντακτών, της Ένωσης των Δημοσιογράφων της Αθήνας, της μεγαλύτερης στη χώρα, ε, είναι άνεργοι. Λοιπόν, πρέπει να βρούμε νέες θέσεις εργασίας. Και τη στιγμή που τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης και κύρια οι εφημερίδες περνάνε μία κρίση και μεταφέρονται σιγά σιγά πολλές διαστηριότητε στο διαδίκτυο, είναι σημαντικό εκεί πέρα η Ευρωπαϊκή Ένωση να θέσει τους κανόνες να δώσει λύσεις. Ε, για την ε, κυρία Καμερέβερ που ξέρω την ε, ιδιαίτερη ανασχόλησή της με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και είναι πολύ σημαντικό και ευελπιστούμε σε μια ανοιχτή επικοινωνία γιατί η ανταλλαγή εμπειριών και προτάσεων μπορεί να χρησιμεύσει στο καλύτερο αποτέλεσμα θέλω να ξέρετε ένα πράγμα θα έχετε την υποστήριξή μας γιατί αναφερθήκατε ε, σε κάτι πολύ σημαντικό. Ναι, είναι βιομηχανία τα μέσα ενημέρωσης, αλλά δεν είναι μόνο βιομηχανία. Φαίνεται και από τον συντελεστή που υπάρχει, άμα εξετάσετε τον αριθμό των απασχολούμενων στα οπτικοακουστικά σαν ποσοστό του ευρωπαϊκού πληθυσμού με το ποσοστό του ακαθάριστου προϊόντος που παράγεται στα ε, οπτικοακουστικά μέσα, θα δείτε ότι υπάρχει ένας σημαντικός πολλαπλασιαστής. Λοιπόν, ε, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, δεν είναι μόνο βιομηχανία. Δεν είναι μόνο βιομηχανία γιατί σφραγίζεις, επηρεάζεις, καθορίζεις τις εξελίξεις, την ταυτότητα, ειδικά στους νέους ανθρώπους. Λοιπόν, να είσαστε σίγουροι ότι θα έχετε την πλήρη υποστήριξη στο Ευρωκοινοβούλιο. Πιστεύουμε ότι θέλουμε, θέλουμε να κινηθούμε μαζί. Και μετά από τις εκτενείς συζητήσεις και διαβουλεύσεις που γίνονται εδώ πέρα, καταλήγουμε, καταλήγεται και ε, γινόμαστε κοινωνοί των, των καλύτερων συνδυασμών, των καλύτερων αποτελεσμάτων. Ε, η, κυρία Κώστα, ε, την ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά της λόγια και συμμεριζόμαστε απόλυτα το ενδιαφέρον σας για τους ανηλίκους. Ε, θεωρούμε ότι η διάσκεψη αυτή που θα διοργανωθεί στην Αθήνα ε, μπορεί και πρέπει να δώσει λύσεις γιατί ξέρετε βρήκαμε, πάνω που βρήκαμε κάποιες λύσεις για την προστασία των ανηλίκων στην ε, τηλεόραση ε, τότε η τεχνολογία προχώρησε ακόμα παραπέρα και έπρεπε να πρέπει να βρούμε γιατί στην τηλεόραση βάζεις ένα σήμα ή βάζεις μια φραγή σε ένα πρόγραμμα αλλά στο διαδίκτυο δεν είναι το ίδιο. Το διαδίκτυο τα παιδιά είναι βάλωτα, τρομερά και Έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα σε όλες τις χώρες. Λοιπόν, πρέπει να βρούμε τον τρόπο να προστατέψουμε το μέλλον της Ευρώπης, γιατί πάνω από όλα αυτό είναι τα παιδιά. Είναι το μέλλον της Ευρώπης. Ε, σε ό,τι αφορά τα θέματα ψηφιοποίησης κλιματογραφικών αρχείων, δεν είμαι ο καθήλυνα αρμόδιος, αλλά θέλω να σας πω και μια άλλη λεπτομέρεια. Ένας τεράστιος πλούτος είναι τα αρχεία των τοπικών εφημερίδων, των μικρών εφημερίδων. Στην Ελλάδα έχουμε εφημερίδες από τις αρχές του 20ου αιώνα και προχωράμε στην ε, ψηφιοποίηση ενός πολύτιμου αρχείου και με τη βοήθεια των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης διασώζεται ένας πλούτος μεγάλος. Ε, για την ε, κυρία Τρούπελ θα συμφωνήσω ότι πρέπει να υπάρχει πολιτιστική ποικιλομορφία Πρέπει, αν θέλετε, αυτό είναι ο πλούτος της Ευρώπης και αυτό είναι που πρέπει να αντιπαραθέσουμε σε μια, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, στην αμερικανική ομογενοποίηση. Ε, δεν είμαστε ίσοι, αλλά δεν είμαστε ίδιοι. Έχουμε όλοι να μάθουμε να προσφέρουμε ο ένας τον άλλον και η, η Ευρώπη πάνω απ' όλα πρέπει να κρατήσει αυτή την πολιτιστική ποικιλομορφία της και δεν υπάρχει Κανένα χώρο πιο σημαντικός για να επιδειχθεί αυτή η ποικιλομορφία από ότι είναι τα μέσα ενημέρωσης. Ε, και τέλος ε, στον ε, αγαπητό πραγματικά κύριο Αγκουράκη, σας εκτιμώ ιδιαίτερα από όλη σα την πορεία στην πολιτική σκηνή, αντίθετα ε, παρά τις πολιτικές μας αντιθέσεις. Ε, δεν δέχομαι ότι δεν υπάρχει ελευθερία έκφραση στα μέσα μαζική ενημέρωση, κύριε Αγκουράκη. Δηλαδή, αν μη τι άλλο, δέστε τα πυρά <laughs> που δεχόμαστε. Ε, υπάρχει, υπάρχουν εφημερίδες, υπάρχουν sites, υπάρχουν... Υπάρχει ελευθερία έκφρασης, υπάρχει. Αυτό που πρέπει να αντιμετωπίσουμε είναι την κρίση στα μέσα ενημέρωσης. Γιατί ξέρετε κάτι, λέτε ότι οι εργαζόμενοι δεν έχουν άποψη, οι εργαζόμενοι πρέπει να προστατευτούν, όμως δεν μπορούν ξέρετε, υπάρχει προϋπόθεση της ύπαρξης του εργαζομένου, είναι η ύπαρξη του εργοδότη. Ε, δυστυχώς η, ζωή αποδεικνύει το άλλο. Είδατε πόσες επιχειρήσεις κλείσανε και πόσοι άνθρωποι μείνανε στο δρόμο. Ε, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να, να, φτιάξουμε το σωστό πλαίσιο. Ε, δεν, ε, σε ό,τι αφορά το επίπεδο των εκπομπών της ιδιωτικής τηλεόρασης και όχι μόνο θα συμφωνήσω μαζί σας, αλλά όταν κάτι το θέλει το κοινό, δεν μπορείς να το στερήσεις. Αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να διαπαιδαγωγήσεις. Και ιδιαίτερα στον χώρο των νέων και ιδιαίτερα με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών μπορούμε να ξεφύγουμε από παγίδες του παρελθόντος. Δεν δέχομαι όμως ότι υπάρχει πλήση εγκεφάλου. Ε, δεν... Ε, δεν δέχομαι ότι, ε, γίνε, ότι υπάρχουν απαγορευμένες απόψεις. Ε, εσείς ο ίδιος είσαστε η διάψευση των όσων λέτε. Σε ένα βήμα με διεθνή προβολή έχετε την ευκαιρία και εσείς και όποιος άλλος έχει αντίστοιχες ή ανάλογες θέσεις ή διαφωνεί. Αυτό είναι δημοκρατία. Λοιπόν, ε, και επειδή αναφερθήκατε και στην περίπτωση της ΕΡΤ και επειδή γνωρίζω ότι υπήρξε εδώ στην Επιτροπή σας εκτενή συζήτηση για το ζήτημα, θέλω απλώς να σας πω δύο λόγια, γιατί σήμερα η δημόσια τηλεόραση λειτουργεί. Σήμερα υπάρχει δημόσια τηλεόραση, δημόσιο ραδιόφωνο με κατοχυρωμένη δια νόμου την ανεξαρτησία της, μπορώ να σας παρουσιάσω και εκτενέστερα στοιχεία για το πώς είναι πλήρως κατοχυρωμένη. Καμία κυβέρνηση ποτέ στην Ελλάδα δεν θα μπορέσει ξανά να επηρεάσει την δημόσια τηλεόραση και αυτό είναι δια νόμου κατοχυρωμένο. Λοιπόν, ε, θέλω απλώς να σας πω, γιατί ήταν μια πολύ δύσκολη απόφαση, μια απόφαση που μπορεί σε εσά εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο να φάνηκε ε, αρνητική. Ε, θέλω να σας πω όμως κάτι, να σας, να σας πω μια προσωπική μου μαρτυρία. Ε, θα σας πω μόνο μια περίπτωση για να δείτε γιατί ήταν ένα οικοδόμημα με πλήρη αδιαφάνεια όπου γινόταν διασπάθηση του δημοσίου χρήματος και δεν υπήρχε καμία δυνατότητα ελέγχου. Θα σας πω ένα παράδειγμα μόνο το, την περίοδο που ήμουν βουλευτής της αντιπολίτευσης και αρμόδιος τομεάρχης για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ε, είχα ασκήσει δρυμύτατη κριτική για ένα σκάνδαλο, απίστευτο σκάνδαλο, ειδικά για την Ελλάδα της κρίσης και μιλάω για τα δικαιώματα του Champions League. Είχε βρεθεί τότε η δημόσια τηλεόραση να προσφέρει 33 εκατομμύρια ευρώ για τρία χρόνια μεταδόσεων τη στιγμή που η επόμενη προσφορά ήταν κάτω από τα 6 εκατομμύρια. Πέντε φορές πάνω είχε δώσει η δημόσια τηλεόραση. Τελείως παράλογο, τελείως εξωφρενικό, τελείως απαράδεκτο για μια χώρα που αιμορραγούσε. Μόλις ανέλαβα την κυβερνητική αρμοδιότητα του χώρου, η πρώτη μου ε, οδηγία ήταν ότι αυτή η σκανδαλώδη σύμβαση πρέπει να λυθεί, πρέπει να καταγγελθεί. Μου υπόθηκε αρμοδίως ότι αυτό είναι αδύνατο γιατί θα πρέπει να το εισηγηθεί η νομική υπηρεσία. Ε, να το εισηγηθεί τότε η νομική υπηρεσία, αφού είναι καραμπινά το σκάνδαλο. Όχι, δεν γίνεται να το εισηγηθεί η νομική υπηρεσία, γιατί είναι η ίδια νομική υπηρεσία η οποία εισηγήθηκε την υπογραφή αυτή τη σύμβαση. Και όταν είπα τότε να αλλάξει η νομική υπηρεσία, γιατί αυτοί οι άνθρωποι προφανώ δεν προφύλαξαν το δημόσιο συμφέρον. Ήταν αδύνατη η απομάκρυνση τη ε, νομική υπηρεσία, η αντικατάστασή τη, γιατί είχαν ισόβιες συμβάσει χωρίς όριο ηλικίας. Ο επικεφαλής της νομικής υπηρεσίας ήταν κοντά στα 80 αλλά δεν μπορούσε να απομακρυνθεί. Λοιπόν, μπορείτε να φανταστείτε ε, αυτό θα το αφήνατε έτσι. Και ήταν μόνο η κορυφή του παγόβουνου το σκάνδαλο του Champions League. Λοιπόν, δεν ήταν. Ήταν μια πολύ δύσκολη απόφαση, σας διαβεβαιώνω. Αλλά μετά από ένα χρόνο προσπαθειών μεταρρύθμισης αναδιάρθρωσης εν λειτουργία αποδείχθηκε ότι αυτό ήταν αδύνατο. Δεν, δεν θέλαμε και δεν είμαστε υπεύθυνοι για το μαύρο γιατί ξέρω ότι κατηγορήθηκε η κυβέρνηση και γι' αυτό το μαύρο έπεσε λόγω της παράνομης κατάληψης του ραδιομεγάρου. Οι μεταδόσεις θα είχαν αρχίσει πολύ πιο σύντομα ε, εάν δεν υπήρχε κατάληψη του ραδιομεγάρου άρχισαν πολύ σύντομα με εναλλακτικά μέσα τώρα απελευθερώθηκε και το ραδιομέγαρο και γίνεται κανονικά η δουλειά στείνεται σε σωστά σε υγιή θεμέλια μια δημόσια ραδιοτηλεόραση πλήρως ανεξάρτητη πλήρως ανταποδοτική που να προσφέρει στους Έλληνες την ενημέρωση αλλά και τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία που δικαιούνται οι Έλληνες πολίτες όπως και κάθε Ευρωπαίος πολίτης. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν θέλουμε να ανοίξουμε παλιές συζητήσεις. Ε, ίσως ήταν ατυχής χειρισμός από την πλευρά σας, ενδεχομένως σήμερα δεν θα κάνατε το ίδιο, αλλά βεβαίως πάντοτε διδάσκεται κανείς από το παρελθόν. Εμείς ε, δεν επιμένουμε, λυθήκαν κάποια προβλήματα και θα ήθελα να ε, ευχηθώ ε, ότι καλύτερο και στην καινούρια και στη νέα δημόσια τηλεόραση. Ε, ας κλείσουμε λοιπόν κάποια θέματα. Εμείς ακούσαμε ότι έχετε πολλές καινούργιες ιδέες. Θέλουμε να σας ευχηθούμε για το επόμενο εξάμεινο κάθε επιτυχία και ελπίζω ε, κάποιοι συνάδελφοι να μπορέσουν. 14-15 Απριλίου δυστυχώς δεν μπορούμε γιατί είναι η τελευταία σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και όλοι όσοι θέλουν να επανεκλεγούν πρέπει οπωσδήποτε να είναι εδώ. Οι άλλοι που δεν θέλουν πάλι θα θέλουν να βρεθούν για τελευταία φορά. Οπότε δύσκολο να βρεθούμε τον Απρίλιο κοντά σας. Ε, πάντως οπωσδήποτε θα έχουμε ευκαιρίες να ξαναβρεθούμε. Σας ευχαριστούμε θερμά και πάλι. Πρόεδρε, if, Μπορώ να στείλω μια πρόσκληση βίντεο προς όλους σας. Γιατί βεβαίως καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν υποχρεώσεις πολλές ε, για τους ευρωβουλευτές, μεγάλες ενηλυμένες υποχρεώσεις. Αλλά θα μπορούσαμε να έχουμε μια βιντεοδιάσκεψη και θέλουμε πάνω απ' όλα προτάσεις σχετικά με το θέμα από εσάς. Γιατί όπως είναι, έχετε την κυρία Κώστα υπάρχουν και, άλλοι, ε, και άλλα μέλη που ασχολήθηκαν πολύ για το θέμα αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Στα διάφορα. Α, έχουμε την το, έγκριση των αποφάσεων των συντονιστών.